ευχηθώ καλή χρονιά και να ευχηθώ καλή χρονιά και στο σύνολο των διερμηνέων που πάντοτε είναι στο πλάι μας με χαρά και καλή διάθεση. Ε, εύχομαι λοιπόν σίγουρα αυτή η συνεδρίαση ε, ξεκινά καλά. Η κυρία Κέλλερ και εγώ εγκαινιάσαμε την ε, γραμμή νυχτερινού τρένου Βιέννης Βρυξελών. Ε, ελπίζουμε ότι τέτοια νυχτερινά τρένα θα δούμε να ε, υπάρχουν παντού και ελπίζουμε κυρία την επόμενη φορά να είστε και εσείς μαζί μας. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης την οποία και εγκρίνουμε αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 6ης Νοεμβρίου και της 3ης Δεκεμβρίου του 19. Εάν δεν έχετε παρατηρήσεις, θεωρούμε ότι ε, εγκρίνονται και στις ανακοινώσεις ε, της Πρόεδρου θέλω να ευχαριστήσω την Γραμματεία για την εργασία της και να ευχηθώ καλή χρονιά. Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε σαν μια ομάδα για να προωθούμε όλα μας ε, τα χαρτοφυλάκια. Ε, σας ευχαριστώ γι' αυτό και πάμε λοιπόν στα, στην έγκριση τύπου για τα οχήματα με ε, κινητήρα, έχουμε τα ελαφρά επιβατικά αυτοκίνητα και εμπορικά αυτοκίνητα, ανταλλαγή πληροφοριών, Euro 5 και Euro 6. Έκθε, ε, εισηγητής μα ο κύριο Βεν Σούλτσε, είναι μια γνωμοδότηση για την αποδοχή των, ε, των οχημάτων, των επιβατηγών αλλά και των ελαφρών επαγγελματικών αυτοκινήτων Euro 5 και Euro 6. Θα σας δώσω χρόνο αγόρευσης για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, κύριε Σιγητά. Έχουμε προθεσμία για υποβολή τροπολογιών στις 29 Ιανουαρίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου. Κύριε Σούλτσε, έχετε το λόγο. Äh, um Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ήδη αναφέρατε το θέμα μας. Εδώ πέρα δεν παίζουμε εμείς τον κύριο Ρολό. Κάνουμε μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή περιβάλλοντος που ασχολείται με το θέμα αυτό της εγκρίσεις τύπων για Euro 5 και Euro 6. Είναι κάπως περίεργο γιατί οι κανόνες αυτοί υπάρχουν ήδη. Υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα το ότι η Κομισιόν τα είχε κάνει τότε στην Επιτροπολογία και υπήρξαν κάποιες ε, καταγγελίες ε, πόλεων ε, και περιφερειών ενώπιον διαφόρων δικαστηρίων. Οπότε η Κομισιόν αποφάσισε τώρα να πάει το θέμα στην τακτική διαδικασία της συναπόφασης, οπότε θα το συζητήσουμε κι εμείς. Ποιο είναι το θέμα μας τώρα. Θα έχετε οπωσδήποτε ακούσει το σκάνδαλο Diesel 2015 περί πειραγμένου λογισμικού που επηρέασε τις εγκρίσεις ε, τύπου. Η Κομισιόν τότε αντέδρασε και εξάδωσε νέους κανόνες και ξαναείδε τα πράγματα στις όριακες τιμές, ε, στα όρια και υπήρξε και ένας παραγόντας συμμόρφωσης γιατί πλέον δεν υπάρχουν μόνο εργαστηριακές ε, μετρήσεις αλλά και ένα μοντέλο το οποίο μετράει τις εκπομπές ε, στον πραγματικό κόσμο. Μεγάλη σημασία εδώ πέρα έχουν τα οξύδια του αζότου, τα οποία ισχύουν μέχρι το 2020 για τα κανονικά γεωταχή. Έχουμε ένα δύο, παράγοντα 2,1, ο οποίος επιβάλλεται για τα κανονικά γεωταχή και ίσως ε, για τα ελαφρά, για τα ελαφρά φορτικά μέχρι το 2021 και τα υπόλοιπα έχουν έναν παράγοντα ένα. Υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να δούμε. Πρόκειται για την ανοχή των ε, φορητών μετρητών, τα όρια ανοχής, ε, που κυμαίνονται στο 0,34. Λοιπόν, αυτά τα οποία σας είπα ισχύουν ήδη στις υπάρχουσες εγκρίσεις ε, τύπου, οπότε θα πρέπει ακριβώς να διορθωθεί το διαδικαστικό λάθος ε, που έχει κάνει η Κομισιόν για μένα δύο ερωτήματα που προέκυψαν σε σχέση με την έκθεση αυτήν. Το ένα είναι εάν ε, θεωρούνται υπεύθυνοι οι κατασκευαστές για αυτό το λάθος ή όχι και εξίσου σημαντικό εάν ε, φταίνε και οι καταναλωτές ε, Σωστό είναι λοιπόν το ότι έκανε αυτή την πρόταση Κομισιόν, αλλά πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι εγώ είμαι κατά, το βλέπετε και στην έκθεσή μου, να υπάρξει μια αλλαγή στους παραγοντές συμμόρφωσης, γιατί είναι θέμα αξιοπιστίας ε, και ασφάλειας δικαίου της Ευρωπαϊκής ε, Νομοθεσίας, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα ε, κινδυνεύσει. Και νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλων ε, να το έχουμε αυτό κατά νου βεβαίως. Δικαίως ε, άλλαξαν ε, οι όριακες τιμές, αλλά το λογικότερο είναι να αναβληθεί αυτή η συζήτηση για τις προδιαγραφές μετά το Euro 6. Εδώ πέρα λοιπόν το σημαντικό είναι να διατηρηθεί η ασφάλεια δικαίου. Έχω μια τροπολογία την οποία θα ήθελα να σας υπενθυμίσω. Είναι τεχνικής φύσης. Η Κομισιόν έχει βάλει αυτούς τους δύο παράγοντες το 1 και το 0,34 ε, σε έναν παράγοντα 1,34 ε, χωρίς να είμαι μηχανικός ρώτησα τη γνώμη των ειδικών και μου είπαν ότι καλό είναι να μείνουν αυτοί οι δύο παράγοντες χωριστά. Ε, είναι ένα τεχνικό ζήτημα και ζητώ την υποστήριξή σας και αναμένω την συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σούλτσου. Κύριε Ντένισον, εσείς έχετε το λόγο εξ ονόματος των σοσιαλδημοκρατών. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, αντικαθιστώ τον Ισμαήλ ο οποίος κολλείεται σήμερα. Όπως είπα, θα ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή. Συμφωνούμε με το ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια σχεδιασμού για τους κατασκευαστές. Υπάρχει και άλλη μια πτυχή ότι η μείωση του παράγοντα συμμόρφωση σε αυτήν την νομοθεσία, όπως λέτε, θα είναι αντιπαραγωγική. Γιατί αν αλλάξουμε τον παράγοντα ο οποίος ισχύει από 1η 2020, θα αμφισβητήσουμε αναδρομικά την ομότητα οχημάτων που έχουν ήδη παραχθεί και καταγραφεί. Και βεβαίως δικαίως υπάρχει η κριτική απέναντι στην αυτοκινητοβιομηχανία. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι παρήγαν τους κινητήρες με βάση τα όσα ήταν νόμιμα την εποχή εκείνη. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ήταν λάθος της Κομισιόν να χρησιμοποιήσει μια πράξη κατηφαρμογή για κάτι το οποίο πιθανότατα απαιτεί την τακτική νομοθετική διαδικασία. Επίσης, ασκήσαμε κριτική στο τεστ ε, πραγματικών συνθήκων οδήγησης που περιέχει ακόμα μεγάλο ποσοστό σφάλματος, το οποίο πρέπει να δούμε γρήγορα. Ε, τούτων λεχθέντων, σας ευχαριστώ και ο Ισμαήλ αναμένει την συνεργασία μαζί σας. Ε, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Φλέγκο για την ομάδα Renew. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή αυτή γνωμοδότηση. Θα ήθελα να πω κάτι ως και ο εισηγητής. Εξ του κόμματος μου. Πέντε χρόνια μετά το σκάνδαλο με τα ντίζελ, οι νέες ε, προδιαγραφές ε, εκπομπών έχουν ε, μειωθεί, αλλά αυτό δεν ισχύει για τα οξύδια του αζότου, τα οποία έκτοτε αυξάνονται. Γνωρίζουμε πόσο βλαπτικές είναι αυτές οι εκπομπές και μεγάλο κομμάτι της ρήπανσης στις ευρωπαϊκές πόλεις οφείλεται ακριβώς ε, στα οχήματα diesel, γύρω στο 30%. Και τα οξίδια του αζότου είναι 66% της ε, ρήπανσης και προκαλούν ε, προβλήματα στην υγεία. Και κοστίζει κιόλας βέβαια αυτό από τη σκοπιά την υγειονομική. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η γνωμοδότηση, χρειάζεται χρόνος για να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπε ο εισηγητής, με τα οποία συμφωνώ. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι αποκλίσεις στις ε, μετρήσεις μεταξύ πραγματικών συνθήκων και εργαστηρίου πρέπει να μειωθούν. Μιλάμε για μεταβατικά μέτρα. Ε, συν το χρόνο με την ανάπτυξη της τεχνολογίας ε, οι αριθμοί αυτοί θα πέσουν. Είναι σημαντικό λοιπόν η Κομισιόν να συνεχίσει την ανάπτυξη του συστήματος μέτρησης σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης για να μην υπάρχουν αυτές οι διαφορές που υπάρχουν σήμερα μεταξύ εργαστηρίου και πραγματικών συνθήκων. Πρέπει λοιπόν να πάμε στην ε, κατεύθυνση των καθαρών αυτοκινήτων, σύμφωνα και με τους στόχους του πράσινου deal. Αλλά χρειάζεται χρόνος ακόμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φλεγκό. Το λόγο έχω εγώ τώρα ως εκπρόσωπος των Πρασίνων γιατί είμαι συνεισηγήτρια για αυτό το θέμα. είναι ένα θέμα που, εκτός του ότι είναι τεχνικό, είναι και πολιτικής φύσης. Και γιατί σας το λέω αυτό. Διότι εγώ έχω διατελέσει αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερεύνης για το Dieselgate. Το σκάνδαλο του Diesel. Πώς φτάσαμε σε αυτή, αυτή την κατάσταση. Ε, δεν θέλω να πιστέψω και ή να εδώ, αυτή την κατάσταση. Έχετε δίκιο κύριε Φλεγκό, έχουμε αυτή την ε, ασθένεια, τη ρήπανση του αέρα που στην Ευρώπη ε, στοιχίζει τη ζωή σε 600.000 ανθρώπους και μέσα σε αυτή τη ρήπανση έχουμε και τα περίφημα οξύδια του αζότου. Έχουμε ασχοληθεί με αυτό και υπάρχουν νέες προδιαγραφές και ακριβώς τι μαθαίνουμε, πως είχε γίνει μια συνεδρίαση ανάμεσα στους ε, υπουργού του περιβάλλοντος στα γρήγορα που είπαν να δεν πειράζει αν δεν μπορείτε να τηρήσετε το ε, προδιαγραφές Ευρώ 6 του 2007, δεν πειράζει, μπορείτε να φτάσετε στο 110% μέχρι το 2020 και μετά 50%, δηλαδή είναι σαν να έχουμε, σαν έχουμε ένα κόκκινο φανάρι μπροστά μας και να, όχι μόνο να μας επιτρέπεται να μην το σεβαστούμε, αλλά και να πατήσουμε και τον γκάζι. Εγώ διαφωνώ με αυτό και πιστεύω πως πρέπει πραγματικά να πούμε πως αυτή η επιτροπολογία έχει λάβει αποφάσεις και κύριε Σούλτσε και εσείς σωστά το αναφέρατε πριν από λίγο, έλαβε αποφάσεις που ήταν ε, υπεράνω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εμείς είμαστε οι εκπρόσωποι των πολιτών και αυτό δεν ελήφθη υπόψη, δεν μας συμβουλεύτηκαν, δεν συμβουλεύτηκαν, ακόμα και το Κοινοβούλιο δεν απέρριψε ε, αυτό το μέτρο. Το ε, πραγματικό ερώτημα είναι όμως πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πέντε χρόνια μετά από το Dieselgate υπάρχουν μελέτες και μάλιστα η τελευταία λέει ότι το νέο μοντέλο diesel εκπέμπει έως και χίλιες φορές περισσότερα μικροσωματίδια όταν να καθαρίζεται το φίλτρο του. Πώς μπορούμε λοιπόν να αφήνουμε αυτή την κατάσταση όταν έχουμε οχήματα που ξεπερνούν όχι μία-δύο φορές πάνω, αλλά χίλιες φορές πάνω. Η Επιτροπή Μεταφορών θα πρέπει να κλείσει τα μάτια μπροστά σε κάτι τέτοιο. Δεν το πιστεύω. Δεν... Έχουμε κράτη-μέλη που δεν σέβονται την οδηγία για τη ρήπανση του αέρα. Υπάρχουν ένα σωρό χώρες που έχουν καταδικαστεί επειδή δεν τη σέβονται. Το θέμα της οδηγίας για την ποιότητα του αέρα. Και εμείς να πούμε, ε, έλα μωρέ δεν πειράζει, είναι ένα τεχνικό θέμα. Όχι, διαφωνώ. Γι' αυτό τον λόγο αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Σιγητά, σας ευχαριστώ πολύ για την εργασία σας. Αλλά πιστεύω πως πρέπει να στείλουμε ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα. Είμαστε νομοθέτες γιατί οι πόλεις καταγγέλουν, γιατί οι πόλεις αποφασίζουν να απαγορέψουν τελείως τα αυτοκίνητα ντίζελ, γιατί κατάλαβαν το εξής, ότι πρώτο με μας μέλημα πρέπει να είναι η υγεία των πολιτών. Εμείς λοιπόν τι θα κάνουμε ως νομοθέτες εάν δεν ε, πάμε προς την κατεύθυνση των πολιτών οι ίδιε οι πόλεις είναι αυτές που θα αναλάβουν τα ενία για αύριο και στη συνέχεια θα μας πούνε μα εσείς η Ευρώπη τι κάνετε τι κάνατε για να μπορέσετε να λύσετε αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο διαφωνώ να μπουν ε, τέτοιοι παράγοντες συμμόρφωσης για τη μέτρηση των ορίων αντοχής γιατί ακριβώς ε, οι κατασκευαστές δεν είναι σε θέση να σεβαστούν ε, προδιαγραφές που ορίστηκαν το 7, δηλαδή 13 χρόνια τώρα. Είναι πολύ απαιτητικέ οι προδιαγραφέ. Δείτε τι γίνεται στι ε, ΗΠΑ ή στην Ιαπωνία. Είναι δύο φορέ πιο απαιτητικέ οι προδιαγραφέ από ό,τι δικέ μα, ειδικά για το οξύδι του αζότου. Μα λέει κανεί λοιπόν ότι δεν, ότι δεν μπορούν να σεβαστούν και να τηρήσουν αυτέ τι προδιαγραφέ. Πιστεύω πω είναι επιτακτική ανάγκη να εγγυηθούμε τον σεβασμό των ορίων του Euro 6 ή στι κανονικέ συνθήκε χρήση και μάλιστα πρέπει να είμαστε κατά και τη ίδια τη αρχή ευελιξία ε, για του ίδιου του κατασκευαστέ. Δεύτερον, πιστεύω πω οι κατασκευαστέ αυτοκινητών θα πρέπει να ε, σχεδιάσουν αυτοκίνητα τα οποία σέβονται τα όρια εκπομπών που ορίζονται από την νομοθεσία. Είναι πραγματικά φρικτό να θυμίζουμε ότι πρέπει να τηρούν τι προδιαγραφέ. Δηλαδή, τι θα πρέπει να κάνουμε, να μην φτιάχνουμε νομοθεσία όσον αφορά τη διατροφή, να πούμε εντάξει μπορείτε να τρώτε δηλαδή ό,τι να και να ξεπερνάτε και τα προδιαγραφέ. Όχι, φέρουμε ευθύνη όσον αφορά τη δημόσια υγεία. Εάν λοιπόν αρχίζουμε να δίνουμε άντε λίγο ακόμα περιθώριο ελιγμού και λίγο περιθώριο ελιγμού, τότε ποια ξεπιστία θα έχουμε εμεί ω νομοθέτε. Δεν είναι φυσιολογικό κάτι τέτοιο. Και τέλο, να πω επίση, γιατί εδώ έχω μια ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ενώ η αγορά αυτοκινήτων, και το βλέπω στη Γερμανία, που είναι πραγματικό ζήτημα, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβλέπει, λέει. Γιατί δεν φτιάχνει ένα σχέδιο εξόδου του ντίζελ, κατάργησης του ντίζελ, ένα πραγματικό πλάνο πρόβλεψης για τα καθαρό αυτοκίνητα. Γιατί υπάρχουν 13 εκατομμύρια κόσμος που δουλεύει στην αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν είναι ούτε στην στον ηλεκτρισμό, ούτε στο υδρογόνο, μα τους ε, ε, Εάν μένουμε με την παλιά τεχνολογία του ντίζελ, αυτό σημαίνει ότι πάμε ε, να χτυπήσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Τι κάνουμε, ναι, λέτε τι γίνεται με το συσσωρευτές, τι θα μας επιτρέψει αυτό να καταρτήσουμε τους ε, υπαλλήλου εφόσον οι, οι ανταγωνιστές μας στην Κίνα ξέρουν πολύ καλά ότι αυτά όλα είναι ξεπερασμένα και εδώ ερχόμαστε και μιλάμε μόνο για συμμόρφωση και για προδιαγραφές. Είναι λογικό αυτό μπορεί να σταθεί. Όχι. Ερώτηση λοιπόν προς την Κομισιόν. Γιατί με αυτό τον κανονισμό για τον ντίζελ που σήμερα ρηπαίνει περισσότερο από την βενζίνη και εδώ θέλω να σας θέσω μια ερώτηση όσον αφορά την τεχνολογική ουδετερότητα, γιατί αυτό μας λέτε συνέχεια. Ε, κύριε Σούλτσε, ε, πιστεύω πως είναι μια γνωμοδότηση που πρέπει να εισακουστεί και έχετε ενστιτοποιήσει το εξή. Πρώτον, τη δημόσια υγεία και δεύτερον, αυτή τον κλάδο. Ξέρω πολύ καλά ότι ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι πολύ σημαντικός στην Γερμανία, όπως και σε άλλες χώρες, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε αυτά τα εκατομμύρια εργαζομένων ε, στην άκρη, γιατί όταν κλείνει ένα εργοστάσιο, στην ουσία κλείνει μια ολόκληρη περιφέρεια και αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να αναγκάσουμε τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να σέβονται τις προδιαγραφές για να είναι Και όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά στο διεθνές ε, επίπεδο. Για την ομάδα ID υπάρχει κάποιος, ο κύριος Μάγερ. Ε, εσείς πήρατε και εσείς το νυχτερινό τρένο. λέγομαι. Ναι, ναι, ήμουνα στο νυχτερινό το τρένο και εγώ. Δεν έχω ε, ουσιαστικά ερώτηση. Είναι γνωστή η κατάσταση. Ευχαριστώ και τον εισηγητή Έχω να πω κάποια πράγματα για αυτά τα οποία είπατε, ειδικά όσον αφορά τον τίτλο. Γνωρίζουμε πως ε, η επιβάρυνση από τα σωματίδια, από την εξάτμιση, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, ε, αυτό το οποίο βγάζει τον ντίζελ είναι καθαρότερο από αυτό το οποίο μπαίνει από μπροστά. Οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη βεβαίω και τους ε, καταναλωτέ και τις ανάγκες ε, της ε, βιομηχανίας όσον αφορά σαφείς κανόνες αλλά και τις θέσει εργασία. Για να βρεθεί μια σωστή ισορροπία νομίζω αυτό είναι προς το συμφέρον όλων. Σας ευχαριστώ. Πίτερ Λουγκεν, έχετε το λόγο. Thank you. Well, it's a little bit of a special day σας ευχαριστώ. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Είναι η πρώτη συνάντηση του έντους, οπότε σκέφτηκα να κάνω κάτι διαφορετικό όπως μια ομιλία στα Όσκαρ. Να ευχαριστήσω τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, αλλά ανταυτού θα ακολουθήσω τη διαδικασία και θα πω ότι στηρίζουμε την πρόταση του εισηγητή να μην αλλάχθούν οι αριθμοί της πρότασης γιατί δεν θα πρέπει ε, να παίζουμε με την επιστήμη και να την δίνουμε μια πολιτική διάσταση. Σας ευχαριστώ η κυρία Κονέτσκα. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφε. Αγαπητοί συνάδελφοι, συντάκτη της γνωμοδότησης, έχω ήδη ξεκαθαρίσει ποια είναι η άποψή μου σε σχέση με αυτήν την έκθεση. Θα ήθελα να πω ότι καλωσορίζω την προσεκτική προσέγγιση ε, του συντάκτη της γνωμοδότησης όπου προσπαθεί να αντιμετωπίσει κάποιους μύθους που συνδέονται με τους παράγοντες συμμόρφωσης. Χαίρομαι που έχει επικρατήσει η λογική των συναισθημάτων. Άρα λοιπόν υποστηρίζω αυτήν την έκθεση. Δεδομένης όμως της έλλειψης νομικής ασφάλειας σε σχέση με τις απαιτήσει για τις μηχανές των ε, οχημάτων και χωρίς να γνωρίζουμε ποιες είναι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την επίδοση, για τις επιδόσεις των οχημάτων. Υποστηρίζω λοιπόν την πρόταση της Κομισιόν χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις και σε ό,τι αφορά την πιο αυστηρή διάσταση και επιβολή των κανονισμών χρειαζόμαστε περισσότερες διευκρινήσεις. Θα πρέπει να υπάρξει έγκριση τύπου όχι μόνο για τους ε, παραγωγούς και τους κατασκευαστές αλλά και για τους ε, καταναλωτές. Χωρίς να γνωρίζουμε τις αποκλήσεις δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Συμπερασματικά θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό το ζήτημα θα πρέπει να συζητηθεί στην νομοθετική διαδικασία αλλά να πούμε και ότι πρόκειται για ένα ζήτημα πολύ τεχνικό που βασίζεται σε επιστήμη και έρευνα και δεν θα πρέπει να είναι πολιτικό ζήτημα. Συνεπώς, στο μέλλον θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσον είναι κατάλληλη η ισχύουσα νομοθεσία ή κατά πόσον χρειάζεται μια πιο βαθιά αλλαγή. Πάντα όμως θα πρέπει να βασιζόμαστε στα στοιχεία και όχι να επηρεαζόμαστε από οποιασδήποτε πιέσεις οι οποίες δεν είναι επωφελείς για μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος άλλο το λόγο? Όχι. Η κυρία Ιωάννα Χισκόφσκα. Non, c'est son Ah, c'est son collègue. Α, είναι κάποιος συνάδελφος. Μάλιστα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο από έξω όνομα της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη γιατί η επικεφαλής της, του τμήματός μας δεν μπόρεσε να βρεθεί εδώ. Βρίσκεται, ε, έχει κάποια άλλη υποχρέωση και δεν μπόρεσε να βρεθεί εδώ σήμερα. Καλωσορίζουμε λοιπόν το σχέδιο γνωμοδότησης του συντάκτη. Θεωρούμε ότι οι περισσότερες προτάσεις μας έχουν γίνει δεκτές και οι τροπολογίες μας φαίνονται λογικές. Θα ήθελα να αναφερθώ μόνο σε ένα ζήτημα. Όταν μιλήσαμε για το Dieselgate, το σκάνδαλο με τα Diesel του 2015, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν εφήρμοζαν τους κανόνες ε, του κανονισμού του 2007. Επρόκειτο λοιπόν για ξεκάθαρη παραβίαση. Αν δούμε τώρα την παρούσα κατάσταση, ε, θα διαπιστώσουμε ότι είναι διαφορετική. Στην ουσία υπάρχει μια νομοθετική πρόταση προς αντικατάσταση ενός κανονισμού, ο οποίος από το Γενικό Δικαστήριο έχει θεωρηθεί ότι ε, δεν είναι κατάλληλος. Δεν έχουμε δηλαδή λανθασμένη εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά αμφισβήτηση του ίδιου του νομοθετήματος. Για λόγους σαφήνειας λοιπόν, η Επιτροπή αποφάσισε να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη νομοθετική διαδικασία έτσι ώστε να εφαρμόσει τους συγκεκριμένους κανόνες. Συμφωνούμε λοιπόν ότι οι οριακές τιμές μπορούν πάντα να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει τώρα όπου το ζήτημα αυτό βρίσκεται σε διάλογο και στόχος φυσικά είναι να υπάρχει νομική ασφάλεια. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρότασή σας για την νομοθεσία κατάργησης των οχημάτων δίζελ, θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε όταν θα συζητήσουμε τα γενικά όρια εκπομπών. Τότε λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρατηρήσή σας και επειδή είναι γνωμοδότηση θα πρέπει να πω ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φτιάξει ένα σχέδιο κατάργηση του ντίζελ για να συνοδεύσει ολόκληρο τον κλάδο μέσω των όσων έλεγε ακριβώς και ο κύριος Σούλτσε πριν γιατί ο κλάδο ε, αντιμετωπίζει σοβαρέ δυσκολίε απέναντι σε παγκόσμιου ανταγωνιστέ. Κύριε Σούλτσε, εγώ θα σα υποβάλω τροπολογία ε, σχετική, γιατί είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση και υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι σε αυτήν. Κύριε Σούλτσε, εσεί ε, τώρα το λόγο για να κλείσετε το θέμα. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για τις παρεμβάσεις σας οι οποίες επιβεβαίωσαν αρκετά από αυτά τα οποία είπα και εγώ και η Κομισιόν. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 29 Ιανουαρίου. Μέχρι στιγμής έχω προγραμματίσει δύο συναντήσεις των σκιωδών, μια τεχνική συνάντηση στις 3 Δευτέρου και μετά στις 17 Δευτέρου που θα συναντηθούμε εμείς θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπατε, κυρία Ντελή. Κάνατε ένα λαθάκι. Μιλήσατε για χίλιες ε, φορές υψηλότερες εκπομπές. Νομίζω ότι αναφέρεστε σε αυτό το οποίο είπε η ΜΚΟ Transport and Environment. Ε, το θέμα όμως αυτό αφορά τον καθαρισμό των ε, καταλητών. Όσοι οδηγούν δίζελ γνωρίζουν ότι μετά από κάποια στιγμή πρέπει να καθαριστεί και ο αριθμός σωματιδίων που βγαίνουν ε, είναι χίλιες φορές ε, ε, μεγαλύτερος σε αυτήν την περίπτωση σε σχέση με την φυσιολογική λειτουργία, έτσι, που στη φυσιολογική λειτουργία είναι σχεδόν μηδενικός. Και Βεβαίω, ε, παρόλα αυτά τηρούν ε, την προδιαγραφή Euro 6, οπότε πρέπει να είμαστε ε, πάρα πολύ προσεκτικοί, μη συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια. Είναι όταν ο καταλήτης βρίσκεται σε λειτουργία καθαρισμού. Αυτό δεν έχει σχέση ε, ουδεμία με το θέμα το οποίο συζητάμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Έχετε δίκιο. Α, είπα, είπα και εγώ ότι είναι όταν καθαρίζονται τα φίλτρα. Ε, ναι, αλλά είναι τότε σε εκείνη τη φάση είναι πάνω από 1000% από το επιτρεπόμενο όριο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε στις τεχνικές συνεδριάσεις, γιατί αν πάρουμε το νούμερο των ε, αυτοκινήτων που δεν σέβονται το ενάγκριστη τύπου Ευρώ 6, είναι 33 εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία κύριε Σόλτσε για αυτό το ενδιαφέρουσα συζήτηση και ελπίζω πως θα ε, τηρήσουμε τις ε, φιλοδοξίες μας. 29 Ιανουαρίου είναι η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Θα εξεταστούν οι τροπολογίες 19 Φεβρουαρίου και η ψηφοφορία στην ε, Επιτροπή μας θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου. Εντάξει, τα σημειώσατε, προχωράμε με το επόμενο σημείο που είναι η διμερή συμφωνία οδικών μεταφορών ανάμεσα στη Γερμανία και την Ελβετία για να εγκριθεί η μεταφορά καμποτάζ σε διεθνείς μεταφορές επιβατών με λεωφορεία και πούλμαν στις διασυνοριακές περιοχές των δύο χωρών. Η συγητής μας είναι ο κύριος Φέρμπερ, αλλά τον αντικαθιστά η κυρία Κέλλερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που μου δώσατε τον λόγο. Αν μου επιτρέπετε το 5 και το 6 θα τα πω μαζί γιατί είναι το ίδιο πράγμα ουσιαστικά εκτός από τις χώρες. Ε, ζητώ συγγνώμη, ο Μάρκους Φέμπερ κολλείται και μου ζήτησε να διαβάσω τα σχόλιά του. Οι δύο αυτές εκθέσεις ε, αφορούν την ε, Γερμανία και την Ιταλία που θέλουν να τροποποιήσουν διμερείς συμφωνίες με την Ελβετία για μεταφορές καμποτάζ στις μεθοριακές περιοχές. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ενέκρινε τη γενική προσέγγιση πέρυσι τον Ιούλιο χωρίς αλλαγές καθώς πρόκειται για τεχνικές εκθέσεις ε, και δεν υπάρχει τίποτα το επίμαχο, υπάρχει μία μόνο τροπολογία που αφορά την νομική βάση για να προσαρμοστεί το κείμενο στη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου και να μην πάμε στον τριμερή διάλογο. Δεν υπάρχουν άλλες τροπολογίες. Ο Μάρκους Φέρμπερ ευχαριστεί τους συναδέλφους για την συνεργασία και προτείνει να υπερψηφίσουμε τις δύο εκθέσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριος Δάνιλσον, εξ ονόματος των Σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Η διαδικασία είναι αρκετά απλή, αλλά το ζήτημα αυτό είναι αρκετά σοβαρό. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελβετίας, Ιταλίας και Γερμανίας έχουν να κάνουν με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Επί της ουσίας συμφωνούμε με την πρόταση του εισηγητή ότι θα πρέπει να δεχτούμε την πρόταση της Επιτροπής και θα σταματήσω εδώ. Κύριε Ετιάν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. For uh, his constructive work on uh, both reports, uh, we would like to welcome. Ε, ευχαριστώ τον Μάρκος για την επικοδομητική του εργασία για αυτές τις δύο εκθέσεις που αφορούν ε, την έγκριση διασυνοριακών ε, γραμμών δημοσίων μεταφορών ανάμεσα στις δύο χώρες. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό λόγω της προσβασιμότητας ε, τα, στην, μετακίνηση με λεωφορεία ή πούλμαν σε αυτές τις διασυνοριακές περιοχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τιέν. Α, και πάλι εγώ είμαι συνεισηγήτρια. Επειδή είμαι πρόεδρος της Επιτροπής, πρέπει να δουλεύω και όλη την ώρα, μάλιστα. Για αυτή την έκθεση πρέπει να σας συγχαρώ, κύριε Φέρμπερ. Προτείνεται κάτι πολύ απλό, μία τροποποίηση απλή, ώστε αυτά τα δύο κείμενα που αφορούν την νομική βάση, λέει ότι πρέπει να διαγραφεί ένα παραπομπή στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της Συνθήκης της Ένωσης. Εγώ πιστεύω πως πρόκειται για μία μη επίμαχη πρόταση που ακριβώς στόχο έχει ε, την, να διευκολύνει τη Γερμανία και την Ιταλία ώστε να διαπραγματευτούν αυτές τις συμφωνίες καμποτάζ για τα λεωφορεία και πούλμαν σε συνεργασία με την Ελβετία. Στηρίζουμε λοιπόν τον εισηγητή και για αυτή τη νομική τροποποίηση που προτείνει. Αυτά. Peter Lundgren, vous ne représentez pas Monsieur Robert Zilleux Κύριε Λόντγκριν, δεν εκπροσωπείτε τον κύριο Ζήλε. Όχι. Ναι, μπορώ, μπορώ. Όχι, δεν νομίζω πως υπάρχει κανένα πρόβλημα εδώ. Το στηρίζουμε. Κυρία Κουντουρά, καλημέρα σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Since ε, Germany... Εφόσον η Γερμανία και η Ιταλία διαπραγματεύονται με την Ελβετία για αυτήν την περιορισμένη εμβέλεια συμφωνία για το καμπατάζ που αφορά τις υπηρεσίες ε, λεωφορείων και ε, πούλμαν, δεν βλέπουμε κανένα λόγο να ε, φέρουμε αντιρρήσεις. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Εξ ονόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποιος θα πάρει το λόγο. Καλημέρα σας κύριε Λιεζουά. Καλή σας χρονιά. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας κυρία Πρόεδρε. Ε, τις θερμότερες ευχές μου επίσης. Ε, καλησπέρα σε όλους και εγώ θα είμαι σύντομος. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Φέρμπερ για την υποστήριξή του και την υποστήριξη προς την πρόταση της Επιτροπής. Όπως σωστά είπατε, η μόνη τροπολογία είναι να αφαιρεθεί μια νομική διάταξη, το άρθρο 2 ένα της συνθήκης και για μας το πιο σημαντικό είναι ότι ε, ε, διορθώνουμε την νομική βάση για τις μεταφορές που είναι το, τις μεταφορές που το άρθρο 31. Κανένα πρόβλημα. Το Συμβούλιο ήδη ανέκρινε την πρώτη ανάγνωση τον Ιούλιο ε, των δύο γραμμών, δηλαδή αφαίρεση του άρθρου 2.1 ως νομική βάση της πρότασης, οπότε βασικά οι δύο θεσμοί βρίσκονται στην ίδια, στο ίδιο πνεύμα που ελπίζουμε σημαίνει ότι θα υιοθετηθεί σύντομα αυτή η πρόταση. Να σημειώσουμε μόνο στο Συμβούλιο, στην πρώτη ανάγνωση, υπήρχαν κάποιες ε, διορθώσεις διατύπωσης, όπου όμως δεν πιστεύουμε ότι θα είναι πρόβλημα για το Κοινοβούλιο ε, και το Συμβούλιο να συμφωνήσουν για αυτές τις μικροαλλαγές και να προχωρήσουν στην γρήγορη υιοθέτηση του κειμένου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λουεζουά και δίνω το λόγο την κυρία Ζελέ. Για να κλείσετε. Μετά από τόσα θετικά δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Παρά μόνο ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και συνεχίζουμε με την απαλλαγή 2018 για το Γενικό Προπολογισμό της Ένωσης. Ε, δύο εκθέσεις έχουμε. Πρώτον αυτήν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έπειτα για τους διάφορους οργανισμούς και κοινοπραξίες στον τομέα των μεταφορών. Επειδή η κυρία Κλάουντια Μοντέρο πρέπει να φτάσει αλλά δεν είναι εδώ ακόμα. Νομίζω πως θα ξεκινήσουμε από τη δεύτερη έκθεση με εσάς κυρία Γκραπίνη για ε, τους οργανισμούς και κοινοπραξίες στον τομέα των μεταφορών. Θυμίζω πάντως ότι ακολουθούμε πάντοτε την ίδια διαδικασία για αυτές τις απαλλαγές των οργανισμών και των κοινοπραξιών ε, και έχουμε έξι ε, οργανισμούς και κοινοπραξίες. Έχουμε το Clean Sky 2, που προσθέθηκε μετά από αίτημα του ΕΛΚ. Έχουμε την ΕΜΖΑ, την ΕΑΖΑ, την ΕΡΑ και τις κοινοπραξίες Caesar, Shift to Rail και Clean Sky. Κυρία Ισηγητρία, λοιπόν, σας δίνω το λόγο για 5 λεπτά για να μας παρουσιάσετε ε, την κατάσταση πρόοδου. Σας ευχαριστω ajutat foarte mult, Σα ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι οι σκιώδει εισηγητέ ήταν μεγάλη βοήθεια, ε, κατέθεσαν τροπολογίες, έχουμε και συμβιβαστικέ προτάσει και να πω εξ αρχή πως εν γέννη τα, οι επιδόσεις των οργανισμών και των κοινοπραξιών το 2018 ήταν θετικές και οι προκλήσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν αυτοί οι οργανισμοί αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία. Όσον αφορά την ΕΜΣΑ, το Μητρό για την για την καταγραφή των κινδύνων ε, ολοκληρώθηκε το 2018 χωρίς ε, κινδύνο ώστε να μην επηρεαστεί το ετήσιο απόθεμα ε, δηλώσεων. Επίσης έχουμε για τον αυτόν τον οργανισμό να εισηγητήσει τους σκιώδεις εισηγητές οι τροπολογίες που κατέθεσαν βελτιώνω το κείμενο και αυτές οι τροπολογίες υπογραμμίζουν το γεγονός ότι ο οργανισμός πρέπει να στηρίξει τα κράτη-μέλη ώστε να μειωθεί ο κίνδυνο στο περιβάλλον στον τομέα της ναυσιπλοείας. καθώς και να καταπολεμηθεί η παράνομη αλία. Τώρα, για την ε, ΕΑΖΑ υπάρχουν συστάσεις όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού που έχει ε, κάνει πολλές ε, προόδους όσον αφορά την ισορροπία των φύλων για να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες υποψήφοι και προσφέροντας ευνοϊκές συνθήκες και ευέλικτα ωράρια για τις άδειε μητρότητας. Έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες, όπως σας είπα, για την ισορροπία φύλων. Έχουμε 17 τροπολογίες που τονίζουν το γεγονός ότι ο οργανισμός θα πρέπει να βελτιώσει τη βιωσιμότητα της αεροπλοείας, να μην ξεχνά γενικά τα θέματα ασφάλειας, αλλά και να εξασφαλίσει ότι λαμβάνει τεχνική βοήθεια εν γέννη για την χρησιμοποίηση των, τη χρήση μάλλον των δεδομένων. Θα πρέπει εδώ να δοθεί περισσότερη ακόμη προσοχή στην ισορροπία των φύλων. Για την οργανισμό για του σιδηροδρόμους τονίζω πως οι δραστηριότητε αυτού του οργανισμού διευρύθηκαν και ε, ως προς αυτό θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να μην υπάρχουν σουκριούσεις συμφερόντων. Ε, νέα καθήκοντα θα ανατεθούν στην ΕΡΑ σύμφωνα με το τέταρτο, την τέταρτη δέσμη για τους σιδηροδρόμους. Η νομοθεσία ε, νέα έχει υιοθετηθεί ως προς αυτό ο οργανισμός έχει ήδη δημοσιεύσει το, τις γραμμέ γραμμές για τη χρήση των ε, ε, σιδηροδρόμων και εδώ έχουμε 17 τροπολογίες και μία συμβιβαστική που αφορά τις μικρομεσαίες. Να μην ξεχνάμε λοιπόν το ρόλο των μικρομεσαίων ε, εφόσον πρόκειται για ορισμό τιμών σας καλώ να υπερψηφίσετε αυτή την τροπολογία, διότι το θέμα των μικρομεσαίων μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές. Χρειάζεται οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες να είναι ανταγωνιστικές και να εξυπηρετούν ολόκληρη την Ένωση. Πρέπει πολλά ακόμα να γίνουν και βεβαίως θα πρέπει να μειωθεί και ο διοικητικός φόρτος σε αυτόν τον τομέα. Τώρα, Σέζαρ, σε, Σέζαρ αυτό η κοινοπραξία έχει δουλέψει για πολλές, πολλούς άξονες, προγράμματα αεροδιαστημικά, γίνεται λόγος για τα ντρόν μέσα στο πλαίσιο του μηχανισμού διασύνδεσης στην Ευρώπη και είναι πολύ θετικό σημαντικό το ότι έχει χορηγηθεί σχετικό κονδύλι. Έχουμε και την, τον γεωγραφικό εντοπισμό, AGS, και επίσης μελλοντική δομή του Ευρωπαϊκού ε, Εναέριου Χώρου. Πρόκειται για διαφορετικά νομικά πλαίσια τα οποία έχουν προσεγγιστεί, ε, αλλά η κατάσταση ακόμα θα εξελιχθεί και είναι αξιόλογο ότι ε, το ΣΕΣΑΡ έχει δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν κατατεθεί 8 τροπολογίες και μία συμβιβαστική που υπογραμμίζει τη δραστηριότητα αυτής της κοινοπραξίας ε, που έχει συμβάλει στην επιτάχυνση των νοτομιών και της χρήσης των τρών στον εναέριο χρόνο και προτείνω να στηρίξετε αυτήν την συμβιβαστική ε, τροπολογία όπου στην ουσία λέγεται ότι τα τρόν θα πρέπει να μπουν σε ένα σύστημα ασφάλειας και εποπτείας αυξημένης πράγμα που σημαίνει και αύξηση του σχετικού κονδυλίου μέσα στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα, όσον αφορά το Shift to Rail, το 2018 σημειώθηκαν σημαντικές πρόοδοι στην ε, εφαρμογή αυτού του ε, προγράμματος Shift to Rail με σημαντικά κονδύλια. Το 2018 οι δράσεις έρευνας και ανάπτυξης σημείωσαν πρόοδο. Όλα λοιπόν βαίνουν καλώς και έχει, έχει μπει σε έναν ε, ε, καλό ρυθμό. Επίσης συνεχίζεται η εφαρμογή της στρατηγικής κατά των απατών για την περίοδο 2017 με 2020. Ήδη φτάσαμε στο 2020. Αυτό σημαίνει ότι καμία περίπτωση αυξημένης παρακολούθησης δεν έχει διαπιστωθεί και άρα Κανένα φάκελο δεν έχει διαβιβαστεί στην Όλαφ. Έχουν κατατεθεί 7 τροπολογίε που μιλούν για την ανάγκη ύπαρξη ενό ενιαίου χώρου σιδηροδρομικών μεταφορών σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα πρέπει να αναζητηθεί δυνατότητα, να αναπτυχθεί αυτή η δυνατότητα μετακίνησης χωρίς εκπομπές και χωρίς ρήπανση είναι σημαντικό αυτός ο τομέας να αποκτήσει περισσότερη ελκυστικότητα και να είναι προσιτός για τους Ευρωπαίους πολίτες. Τώρα, το Clean Sky 2 που είναι η τελευταία κοινοπραξία, να σας πω ότι αυτή η κοινοπραξία θα αναθεωρήσει τον δημοσιονομικό της κανονισμό για να εισάγει νέα πρότυπα και δημοσιονομικές προδιαγραφές σύμφωνα με τον τελευταίο κανονισμό τον 1046. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Δημοσιονομικού Ελέγχου έχει εκδώσει πολύ σημαντική σύσταση για, αυτό, τον, για αυτή την κοινοπραξία με ε, ολοκληρωμένο μητρό ε, κινδύνων. Έχουν διαπιστωθεί μέσα στο 2018 η πρόεδρος διακόπτη. Α, ναι, ναι, ναι, ολοκληρώνω δύο λεπτά. Έχουν κατατεθεί λοιπόν και εδώ τροπολογίες και ε, έχουμε καταφέρει να βρούμε και μία συμβιβαστική η οποία χαιρετίζει τις δραστηριότητες ε, της κοινοπραξίας Clean Sky 2. Σας καλώ να παρακολουθήσετε τις ενδείξεις ψήφου στο κατάλογο ψηφοφορίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γραπίνη. Ξεκινάμε τη συζήτηση. Η κυρία Τάλερ έχει το λόγο. Εξ του ΕΛΚ. Thank you, Chair. Dear um, colleagues, um, Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι υπηρεσίες έκαναν καλά τη δουλειά τους, όμως ε, καθώς ε, πηγαίνουμε προς ένα πιο αποτελεσματικό τομέα μεταφορών πρέπει να έχουν αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια, ειδικά η υπηρεσία σιδηροδρόμων θα χρειαστεί κάθε στήριξη και ίσως και πίεση από το Κοινοβούλιο για να δούμε μια πραγματική ευρωπαϊκή σιδηροδρομική περιοχή, χώρο μέχρι το 2030. Θα ήθελα να τονίσω τρία πράγματα πριν από τις αυριανές ψηφοφορίες. Πρώτον, ε, η μετακίνηση στον σιδηρόδρομο. Η δουλειά η οποία γίνεται από αυτό το εγχείρημα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τους στόχους ε, της πολιτικής μας και αν συγκρίνουμε τον βαθμό αυτοματισμού μεταξύ δρόμων και σιδηροδρόμων βλέπουμε πως υπάρχει κάποιο περιθώριο βελτίωσης. Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί το 2018 είχαμε το σημασία που δόθηκε στα σχετικά προγράμματα στον ορίζοντα 2020. Δεύτερον, θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες ε, όσον αφορά την προκαταβολή των 52 εκατομμυρίων ευρώ της ΕΑΖΑ. Τρίτον, να τονίσω ότι εάν όλα τα αεροπλάνα πετούσαν με τις εφευρέσεις του Clean Sky, θα εξοικονομούσαμε 180 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα ετσίως. Ε, ουσιαστικά πρόκειται για τις εκπομπές ενός ε, μεσαίου κράτους μέλους, ε, π.χ. της Ολλανδίας ενός έτους ή δυόμιση φορές οι εκπομπές της χώρας μου, της Αυστρίας. Έχω υποβάλει μια τροπολογία σχετικά και ελπίζω να την στηρίξετε, γιατί αυτά πρέπει να είναι γνωστά. Είναι ένα τεράστιο επίτευγμα της ευρωπαϊκής έρευνας και ανάπτυξης να τελειώσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τους ε, συναδέλφους, ειδικά την εισηγήτρια, την κυρία Γκραπίνη και βεβαίως προς όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν για ε, ε, τις απαλλαγές αυτές. Ευχαριστώ. Κύριε Έτιεν, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ θα πω και ευχαριστώ στην κυρία Γκραπίνη και στους ε, σκιοδησηγητές. Είχαμε μια αρκετά καλή συνεργασία και όταν υπάρχει καλή συνεργασία έχουμε καλά αποτελέσματα. Και νομίζω ότι 7 λεπτά αντί για 5 για 6 τέτοιε υπηρεσίε ε, δεν είναι υπερβολικό. Δηλαδή, άλλο κόσμο μιλάει 7 λεπτά για άλλα και άλλα. Οπότε καλό είναι να μπαίνουμε στις λεπτομέρειες όταν ε, μιλάμε για την απαλλαγή. Κανονικά οι απαλλαγές είναι τεχνικές και όχι πολιτικές. Καλό είναι όμως να γινόμαστε και πολιτικοί, όπως είπατε και εσείς κυρία Τάλερ. Ε, υπάρχουν πολλές δουλειέ που πρέπει να γίνουν από τη χύψη υπηρεσία, οπότε χρειάζονται λεφτά. Και θα ήθελα να τονίσω ότι ειδικά τα κοινά εγχειρήματα όπου ξοδεύουμε χρήμα των φορολογουμένων, αλλά σε συνεργασία με την βιομηχανία μπορούμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Ειδικά για το πράσινο deal που έχουμε τώρα μπροστά μας, τα εκείνα αυτά εγχειρήματα όπως ο καθαρός ουρανός είναι πολύ επιτυχημένα. Καλοδεχόμενη λοιπόν η τροπολογία σας κυρία Τάλερ για την Ολλανδία παρά το ότι βασίζεται σε στοιχεία του 2015 αν είχαμε πιο επίκαιρα στοιχεία, θα αφορούσαν μια ακόμη μεγαλύτερη χώρα. Μπορείτε να το δείτε. Αλλά το σκεπτικό είναι καλό. Θέλουμε να δείξουμε δηλαδή το τι σημαίνει, γιατί κάνουμε αυτή την έρευνα και ποιο θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμά της ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Να τονίσω ότι η συγγήτρια προσπάθησε να κάνει κάποιες συμβαστικές ε, τροπολογίες ε, για το ERRRA, την ε, τροπολογία 16 του Renew και του ID. Καλό αυτό, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι νομίζω ότι η τροπολογία του Renew είναι καλύτερη. Οπότε αυτήν θα ήθελα να ψηφίσετε και όχι την ε, συμβιβαστική. Αυτά από μένα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τιέν. Κύριε Ρόντο, καλημέρα σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους εισηγητές ε, για τα σχέδια γνωμοδότησης. Τα στοιχεία που ε, παρουσιάστηκαν εδώ στην ουσία εκφράζουν πολύ την άποψή μας. Καλωσορίζουμε το ζήτημα της πρόκλησης της σώτας των φύλων ε, στην ΕΑΖΑ. Επίσης συμφωνούμε με την υιοθέτηση μέτρων για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και επίσης θέλουμε να πούμε ότι θα πρέπει για όλους τους οργανισμούς να έχουμε δικλείδες ασφαλείας για την προστασία από τη σύγκρουση συμφερόντων. Γενικά πιστεύουμε ότι οι γνωμοδοτήσεις απαλλαγής θα μπορούσαν να παρουσιάσουν καλύτερα την έλλειψη προόδου σε ό,τι αφορά την αλλαγή στις μεταφορές και άρα υποστηρίζουμε τις τροπολογίες των συναδέλφων. Επίσης, θα θέλαμε να αναφερθούμε στο ζήτημα της αεροπλοείας. Η έλλειψη φορολογίας στον τομέα των αερομεταφορών στην ουσία σημαίνουν ότι ίσως ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός να έχει οδηγήσει σε υψηλότερες εκπομπές. Το γεγονός ότι αυξάνουμε την αποτελεσματικότητα δεν σημαίνει ότι συνολικά μειώνονται οι εκπομπές. Άρα θεωρούμε ότι στον τομέα των αερομεταφορών εκεί θα πρέπει να κάνουμε επιπλέον δουλειά για να υποστηρίξουμε την συνολική μείωση των εκπομπών. Θεωρώ ότι ίσως το μοναδικό που θα βοηθήσει είναι η αύξηση των φόρων σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φρέοντι για το ID. Δεν υπάρχει κανείς. Η κυρία Ντάλι, εξ ονόματος της ΚΟΕ. Ντέιλι, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα αναφερθώ στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις δικές μας τροπολογίες και ιδίως ε, σε ό,τι αφορά την ΕΑΣΑ. Η δική μας ε, η ομάδα υποστηρίζει ότι θα πρέπει να αυξηθεί το ανθρώπινο δυναμικό και τα οικονομικά μέσα του οργανισμού αυτού έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεί καλύτερα τις αρμοδιότητές του. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι απλά η αύξηση του προπολογισμού δεν είναι λύση, το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά κάποιες φορές η εργασία αυτών των οργανισμών επηρεάζεται από την έλλειψη χρημάτων και από την έλλειψη προϋπολογισμού. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι θα γίνει και έρευνα τώρα για το Boeing ε, MAX 737. Θεωρούμε επίσης ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθούν και τα διοικητικά συμβούλια αυτών των οργανισμών. Σε ό,τι αφορά το Clean Sky, για εμάς το σημαντικό εδώ είναι να εξετάσουμε το πώς μπορούμε να έχουμε μια ξεκάθαρη στρατηγική για την πρόληψη της απάτης. Το 2018 είχαμε σχετικές καταγγελίες και φυσικά έχει υπάρξει ενθουσιασμό σε σχέση με την επιτυχία αυτού του εγχειρήματο από κάποιε ομάδε, αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Όπω είπαν και οι προηγούμενοι ε, ομιλητές θεωρώ ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και να υποστηρίξουμε τις ε, γνωμοδοτήσεις και ανυπομονούμε ε, για τη συζήτηση αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ και στρέφομαι στην Κομισιόν και θα δώσω το λόγο στον κύριο Δεδίος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω την πρόταση γνωμοδότησης σε σχέση με τους ε, οργανισμούς αυτούς και τις κοινέ επιχειρήσεις. Αν υπομονούμε να επιβεβαιωθούν όλα αυτά στην αυριανή ψηφοφορία, σε ό,τι αφορά το αίτημα περαιτέρω πληροφόρησης από το ΕΛΚ, θα μπορέσουμε να σας δώσουμε αυτές τις πληροφορίες αργότερα σήμερα το απόγευμα. Αυτές οι πληροφορίες έχουν να κάνουν με το Shift to Rail και το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες σας αυτές τις ε, παρεμβάσεις. Να θυμίσω ότι η ψηφοφορία θα γίνει αύριο, 21 Ιανουαρίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού θα γίνει στις 19 ή 20 Φεβρουαρίου και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει στη δεύτερη σύνοδο του Μαρτίου. Αλλά αύριο θα ψηφίσουμε εμείς και συνεχίζουμε. Με την κυρία Κλάουντια Μοντέρο. Ε, αλλάξαμε τη σειρά γιατί δεν είχατε φτάσει ακόμα. Ε, έχετε το λόγο σε σχέση με την απαλλαγή για το 2018 και ξεκινάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύρια Μοντέρο, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη που αναγκαστήκατε να αλλάξετε την ημερήσια διάταξη γιατί ήμουνα στην Επιτροπή Αλίας όπου εκεί ε, έχω αναλάβει έναν άλλον φάκελο που έχει να κάνει με την Αλία. Σε ό,τι αφορά τώρα την έκθεση που συζητάμε εδώ. Είναι ξεκάθαρο ότι πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που παρουσίασαν τις τροπολογίες. Έχουμε σύνολο 22 τροπολογίες και ε, δύο συμβαστικές ε, τροπολογίες. Και τώρα θα εστιάσω περισσότερες τροπολογίες γιατί μπαίνουμε στην ουσία στα βασικά θέματα αυτής της πρότασης. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 6, οι συντονιστές θα παρουσιάσουν τα αιτήσιους λογαριασμού στο Κοινοβούλιο και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει αυτό το θέμα να συζητηθεί σε ένα άλλο φόρουμ και όχι εδώ. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 15 για την τροποποίηση του συστήματος του προϋπολογισμού. Επίσης δεν θα πρέπει να συζητηθεί τώρα, γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο είναι αρκετά ασαφές. Να πω επίσης ότι θα ψηφίσω θετικά τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τις νέες υποδομές συντήρησης και ασφάλειας ε, των ε, υπαρχόντων υποδομών, των υπαρχουσών συγγνώμη, υποδομών. Επίσης, τροπολογίες που έχουν να κάνουν ε, με τα δικαιώματα των επιβατών, τον βιώσιμο τουρισμό και την εκτέλεση των διαρθρωτικών ταμείων και μεδεντικών ταμείων. Για όλα αυτά θα ψηφίσω θετικά. Γνωρίζουμε επίσης ότι έχει γίνει μια τροπολογία ε, ότι έχει γίνει μια τροπολογία η οποία έχει να κάνει με την ανταπόκριση σε περιπτώσεις ανθρωπιστικής κρίσης ή και φυσικών καταστροφών. Αυτές οι τροπολογίες λοιπόν έχουν κατατεθεί και εφόσον έχετε κάποια, κάποιο ερώτημα σε σχέση με όλα αυτά, μπορείτε να με ρωτήσετε, να μου απευθύνετε τις ερωτήσεις σας. Δεν έχω ακούσει όλη τη συζήτηση, ήμουνα στην Επιτροπή Αλίας, οπότε αν υπάρχει κάποια άλλη τροπολογία που θέλετε να κάνετε, είμαι δύο στη διάθεσή σας για να με την παρουσιάσετε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μοντέιρα. Κυρία Γκραπίνη, έχετε δύο λεπτά. Εξ ονόματο των Σοσιαλδημοκρατών. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Η ομάδα μου ανέλησε το κείμενο Έχουμε επίσης αναλύσει τις συμβιβαστικέ και συμφωνούμε με τις συμβιβαστικέ που πρότεινε η συγγήτρια. Νομίζω πως αυτές οι δύο συμβιβαστικέ καλύπτουν πάρα πολλά πράγματα και πιστεύω πως αύριο θα έχουμε ένα ε, ενωπημένο κείμενο που θα υπερψηφιστεί. Μετά από την παρέμβαση της Κομισιόν στις άλλες εκθέσεις δεν είχα την ευκαιρία να παρέμβω όμως κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να απαντήσω σε δύο συναδέλφους για τις απαλλαγές. Καταρχάς η πρόταση του Ρινιού συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο της συμβιβαστική τροπολογίας. Δεν υπάρχει καθόλου λοιπόν ε, ε, όπως είπα, διαφοροποίηση της πρότασης, με την οποία εξάλλου συμφωνώ. Έπειτα, πιστεύω πως δεν έπρεπε να κατονομάσουμε κάποια χώρα σε τροπολογία, γι' αυτό και δεν συμφώνησα ε, να κατονομαστεί χώρα. Δεν νομίζω πως είναι καλό το να κάνουμε κάτι τέτοιο, κυρίως γιατί τα δεδομένα τα οποία αναφέρονται δεν είναι ενήμερα. Και γι' αυτό και δεν ήθελα να στηρίξουμε αυτή την τροπολογία, διότι, όπως σας είπα, αναφερόταν ονομαστικά μια χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γραπίνη. Κύριε Τιέν, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους του κυρίου Μπάουσα Ντίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μοντέιρο για την πολύ επικοδομητική της προσέγγιση σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, θα ήθελα να αναφερθώ στις καθυστερήσεις που έχουν υπάρξει και θα ήθελα να προσκαλέσω τους συντονιστές να επιταχύνουν τη διαδικασία σε σχέση με τους διαδρόμους των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Κομισιόν να προτείνει ένα νέο μηχανισμό που προσανατολίζεται προς τα αποτελέσματα με σχεδιασμό μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο έτσι ώστε να φτάσουμε στους στόχους μας. Σε ό,τι αφορά την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, θα πρέπει να επιτύχουμε τους στόχους της ψηφιοποίησης και της ασφάλειας και άρα χρειάζεται καλύτερο συντονισμό των προγραμμάτων εργασίας έτσι ώστε να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ε, τομέων της ενέργειας, των μεταφορών και ε, του, τον ψηφιακό τομέα. Τρίτον, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. Και σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ECA, πολλοί επιβάτες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και δεν μπορούν να επωφεληθούν από την προστασία αυτή. Άρα θα πρέπει να ε, ενισχύσουμε το πλαίσιο των δικαιωμάτων ε, των επιβατών ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει επίσης μεγάλη ευκαιρία να δημιουργηθούν συνέργειες ανάμεσα στα διάφορα δίκτυα μεταφορών και άρα ο τομέα τη στρατιωτική κινητικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την πολιτική μα για τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Ε, αυτό θα μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε σε φυσικές καταστροφές ε, καθώς και ανθρωπιστικές κρίσεις. Εκ μέρους του κυρίου Μπάου Σαντίας θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μοντέρο για ακόμα μια φορά για την στήριξή της και τη συνεργασία της. Ευχαριστώ. Uh, uh. ε, ευχαριστώ Πρόεδρε εκ μέρους των Πρασίνων, όπως είπαμε και τον Δεκέμβριο, εμείς δεν θέλουμε να δοθεί μια στρατιωτική διάσταση στο Connecting Europe και άρα δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί αυτή η διάταξη για τις στρατιωτικές μεταφορές. Στο κύριε Φρόντ. Κύριε Ντέλη, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι επίμαχες οι διαδικασίε ή τροπολογίε οι περισσότερες και μπορούμε να τι ρίξουμε. Βεβαίω το παραπάνω μα είναι η προσθήκη της στρατιωτικής κινητικότητας ε, στο διευρωπαϊκό δίκτυο ε, μεταφορών και η πρόταση της ε, Κομισιόν ε, για μια χρηματοδότηση 6,5 εκατομμυρίων. Κοιτάξτε, αν λέμε ότι χρειάζονται αυτά τα λεφτά για φυσικές καταστροφές και ανθρωπιστικές κρίσεις, καλύτερα να τα ξοδεύαμε αντιμετωπίζοντας ζητήματα κλιματικής αλλαγής που προκαλούν πολλές από τις καταστροφές που δεν είναι φυσικές ε, αλλά προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. Και δεν θα χρειαζόταν ανθρωπιστικές παρεμβάσεις αν δεν ξοδεύαμε τόσα λεφτά σε στρατιωτικοποίηση και παρεμβαίναμε σε άλλες χώρες. Αλλά σε γενικές γραμμές ε, το στηρίζουμε και είμαστε υπέρ της διαγραφής ε, του συγκεκριμένου. Ε, συνολικά όμως θέλουμε να τονίσουμε την σημασία μιας πιο ποιοτική ανάλυσης και οπωσδήποτε είμαστε υπέρ της τροπολογίας αυτής που υπενθυμίζει στην Κομισιόν ότι δεν είναι το μόνο κριτήριο απόδοσης ε, το ποσό των χρημάτων που ξοδεύεται και θέλουμε να το δει πιο εις βάθος η Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Αυτή η Κομισιόν δεν θέλει κάποιος. Θυμίζω λοιπόν ότι η ψηφοφορία θα γίνει αύριο, 21 Ιανουαρίου, η ψηφοφορία στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού θα γίνει 19 και 20 Φεβρουαρίου και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα είναι για τη δεύτερη σύνοδο του Μαρτίου. Και συνεχίζουμε με την, για ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μάθιου Μπόλτουιν που είναι ο Ευρωπαίος Συντονιστής για την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές. Φτάνει. bonjour, bienvenue dans notre commission. Bonne année à vous. Καλώ ήρθατε. Καλή χρονιά έχει σε εσά. Και έχουμε τη χαρά να σας υποδεχτούμε. Ευχαριστούμε που απαντήσατε στην πρόσκλησή μας και που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας. Ξέρετε ότι ο στόχος αυτής της επίσκεψης είναι να γίνει μία ει βάθο ανταλλαγή απόψεων για αυτή τη στρατηγική, την περίφημη στρατηγική πού βρισκόμαστε όσον αφορά την πρόοδό και τις ε, δράσεις σε κλειδιά. Η ασφάλεια η οδική έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες και η ευρωπαϊκή δρόμη είναι η ασφαλέστερη στον κόσμο. Δυστυχώς ο αριθμός των ε, νεκρών και των τραυματιών παραμένει υψηλός και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οθετήσει μια προσέγγιση, την προσέγγιση της ορατότητας μηδέν του ασφαλού συστήματος για να αποφευθούν οι σοβαροί τραυματισμοί στους δρόμους. Αν τα νούμερα είναι ακριβή, δηλαδή ένας θάνατος ισοδυναμεί με 7 σοβαρούς τραυματίες στους δρόμους. Χρειάζεται λοιπόν πραγματικό συντονισμό με το Κοινοβούλιο, τα κρατημέλη αλλά και τις πόλεις και όλους τους φορείς που ε, ασχολούνται με την ε, ασφάλεια, την οδική ασφάλεια. Σε συγχαίρω λοιπόν για τη δουλειά σας που δεν αναγνωρίζω. Γνωρίζετε επαρκώ, ενώ πρόκειται ε, για ένα τομέα σημαντική δράση και επίση για το ότι δίνεται σημασία σε έναν τομέα που μας ενδιαφέρει ειδικά όταν μιλάμε για βιώσιμη κινητικότητα με τη βοήθεια συστημάτων, ε, φιών συστημάτων ή των ε, μικρών εκπομπών. Κυρίως όμως θέλουμε να στείλουμε ένα σχηρό μήνυμα για προστασία των χρηστών των ε, δρόμων και κυρίως των πιο ευάλωτων, δηλαδή των ποδηλατών ή των πεζών. Ε, πρώτα λοιπόν θα δώσω το λόγο σε εσά για να μας ε, πείτε ακριβώς πού βρισκόμαστε, πράγμα που μετά θα μας δώσει λαβή για ερωτήσεις. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντέλη και ευχαριστώ για τα πολύτιμά σας και κέρια σχόλια. Θα προτιμήσω να μιλήσω όμως τώρα στην ε, μετρική μου γλώσσα. Καλησπέρα σας. Ε, Κυρίε και κύριοι, είναι μεγάλη μου τιμή που με καλέσατε για να μιλήσω για δύο θέματα που ε, σας απασχολούν ιδιαίτερα, όπως είπατε, την οδική ασφάλεια και την ε, βιώσιμη μετακίνηση. Παραμένω Γενικός Διευθυντής στην Γενική Διεύθυνση μου, αλλά μου ανατέθηκε και αυτός ο νέος ρόλος Ευρωπαίος της Οδικής Ασφάλειας. Και το έκανα με ιδιαίτερη μου χαρά γιατί η οδική ασφαλεία ε, παραμένει ένα βασικό ζήτημα που δεν έχει επιληθεί στην Ευρώπη και παγκοσμίω και είναι και προσωπικό μου πάθος και σχετίζεται και με την ε, ε, βιώσιμη κινητικότητα όταν έχουμε παραδείγματος χάρη καλύτερες υποδομές για πεζούς και ποδηλάτες, δίνουμε και κίνητρα και κάνουμε τη μετακίνηση αυτή πιο ασφαλή. Καθώς λοιπόν η πυρος γίνεται πιο αστική, 80% κατά το 2050 υπολογίζεται, να έχει μεγαλύτερη σημασία η οδική ασφάλεια και ε, οι ευπαθείς ε, επαχούμενοι, δηλαδή ποδηλάτες και μοτοσκλήτσες κλπ, είναι 70% των θυμάτων. Το κόστος είναι γύρω στο 3 ε, εκατομμύριο ευρώ το οποίο υπολογίζεται σε ρήπανση αλλά και κυκλοφοριακή συμφόρηση και τα σχετικά. Πρέπει λοιπόν να δούμε τις πολιτικές που θα μειώσουν όλο αυτό το εξωτερικό κόστος, όπως να μειωθεί η εξάρτησή μας από κινητήρες ε, εσωτερικής καύσης της πόλης. Βεβαίω αυτό μας οδηγεί σε μια λεπτομερή στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε τις εκπομπές στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Deal ε, που ξέρω ότι θα συζητήσετε με την Επίτροπο και τον επόμενο μήνα και στην Ολομέλεια στις 29 του μηνός. Να ξεκινήσω λοιπόν με την οδική ασφαλεία και την έκταση του προβλήματος. Ε, λοιπόν, θα μιλήσω λίγο γρήγορα, γιατί ξέρω τα γνωρίζετε. Οι αριθμοί αυτοί, τους οποίους ξέρετε πολύ καλά, είναι απλά απαράδεκτοι. Είναι μια λέξη πολύ χρησιμοποιημένη και τη χρησιμοποιώ, αλλά το περίεργο είναι ότι τους δεχόμαστε τελικά. Δηλαδή αν δούμε το τι γίνεται στην αεροπορία παραδείγματο χάρη, δεν θα το δεχόμασταν ποτέ να έχουμε τέτοιους αριθμούς ε, νεκρών. Και λέμε ε, ότι πρόκειται για ατυχήματα, σε ε, να ήταν δηλαδή κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Και σας παρακαλώ να θυμάστε ότι αυτά συμβαίνουν σε δημόσιο χώρο. Δηλαδή πρέπει κάπου να αναγνωρίσουμε ότι εμείς οι δημόσιες αρχές κάτι δεν κάνουμε όσον αφορά την ευθύνη μας για να είναι ασφαλής η ανθρωπική Και η πραγματικότητα είναι ότι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε επιτέλους. Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι της οδικής ασφαλής είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Έχουμε κάποιο ιστορικό, το οποίο βλέπετε εδώ πέρα. Καθορίσαμε για πρώτη φορά στόχους το 2001. Τα καταφέραμε την πρώτη δεκαετία, μειώθηκαν οι θάνατοι κατά 43%. Δεν τα καταφέραμε στη δεύτερη δεκαετία. Μειώθηκαν μόνο κατά 21% ενώ ο στόχος ήταν 50%. Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερος ε, για το ότι οι Υπουργοί Μεταφορών στην Βαλέτα επαναβεβαίωσαν τον στόχο του 50% για την επόμενη δεκαετία μέχρι το 2030 και για πρώτη φορά ε, να περιλάβει αυτό και τους σοβαρούς τραυματισμούς. Είδω λοιπόν τι γίνεται ναι, αν το δούμε από το υψηλότερο σημείο του 1972 όταν είχαμε 200 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων φτάσαμε στο 2015 σε 50 θανάτους ανά εκατομμύριο και βλέπετε οι τελείες είναι η απόδοση του κάθε κράτους και βλέπετε ότι έχει μειωθεί και η απόκληση μεταξύ των κρατών μελών αλλά σημειώστε επίσης στα δεξιά βλέπετε πως κάποια στιγμή έχει κολλήσει από το 2013 και δεν μειώνεται άλλο. Εδώ πέρα βλέπετε την άκρη αυτού του διαγράμματος, είμαστε στο 2010 και μετά ουσιαστικά είναι ευθεία γραμμή. Αν δει κανεί λοιπόν τις λεπτομέρειες τα χρόνια μέχρι το 2010, οι θανάτοι επιβατών έχουν μειωθεί κατά 26%, πεζών κατά 17%, μοτοσυκλωτιστές κατά 16%, ποδηλάτες κατά 5%. Ο αριθμός λοιπόν των ευπαθών χρηστών του δρόμου πλέον έχει ίδιο αριθμό θανάτων με τους επιβάτες. Οπωσδήποτε λοιπόν έχουν γίνει τα πράγματα πολύ πιο ασφαλή για τους επιβαίνοντες στα αυτοκίνητα, αλλά όχι για αυτούς που είναι έξω από τα αυτοκίνητα. Εδώ λοιπόν βλέπετε το πώς θα κάνει η δική σας η χώρα, αλλά βεβαίως δεν μπορείτε να δείτε ποια είναι η χώρα σας από τόσο μακριά. Στα αριστερά είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Σημειώστε επίσης ότι η Δανία και η Ιρλανδία επίσης είχαν σημαντική μείωση. Αλλά υπάρχουν δύο χώρες, Σουηδία και Ολλανδία, που ιστορικά τα πήγαιναν πάρα πολύ καλά, που έχουν αύξηση. Στα δεξιά είναι οι χώρες που φέρνουν περισσότερο. Αν δείτε ε, τα διαγράμματα βλέπετε ότι γίνεται μεγάλη πρόοδος, αλλά υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει ακόμα. Και κάπου εκεί, τέρμα δεξιά, αν δούμε την ευρύτερη Ευρώπη, ε, η καλύτερη χώρα είναι η Νορβηγία. Και το Όσλο, το οποίο λαμβάνει ριζικά μέτρα τα τελευταία χρόνια, είχε έναν θάνατο αποτροχαίο το 2019 και ε, μηδέν θανάτους ευπαθών χριστών. Ε, κανέναν θάνατο παιδιών κάτω των 15. Οπότε όταν λέμε ότι είναι κάτι αδύνατο, ε, μπορεί να γίνει. Σύντομα λοιπόν, αυτά είναι κάποια από τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οδική ασφάλεια. Δεν χρειάζεται τώρα σε εσάς να πω πράγματα για να σας πείσω το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αναφερθώ σε κάποια πράγματα πρώτα απ' όλα στο τέταρτο, στην χρηματοδότηση και να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας γιατί χρηματοδότησε τρία πιλωτικά για την οδική ασφάλεια, κυρίως ε, ένα πρόγραμμα ανταλλαγών ε, προς όφελος έξι χωρών και αύριο θα πάω να συναντήσω κάποιες από αυτές στην ΡΕΝ για να μάθω τι κάνουν οι Γάλλοι. Ξεκινήσαμε επίσης να δούμε τα δεδομένα των αυτοκινήτων και οι μελέτες αυτές είναι κάτι που θα δούμε τον Φεβρουάριο. Πέρσι λοιπόν ορίσαμε μια νέα στρατηγική οδικής ασφάλειας η οποία αναπτύχθηκε τον Ιούνιο του 2018 σε ένα έγγραφο εργασία ε, για να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η στρατηγική. Όχι μόνο νομοθετική, αν και δεν φοβόμαστε βέβαια να νομοθετήσουμε, ε, με την βοήθειά σας. Ε, πέρσι το κάναμε και για την ασφάλεια των οχημάτων και των υποδομών και προχωράμε γρήγορα. Μιλάμε και για το τι προσπαθούμε να πετύχουμε σε σχέση με κάποιους ε, μετρήσιμους δείκτες. Εάν δεν μετράμε δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Και συμφωνήσαμε λοιπόν με τα κράτη-μέλη να συλλέγουμε δεδομένα στους εξής 8 ε, τομείς. Θα τα μετράμε από το 2020 και θα έχουμε έτσι μια αίσθηση του ποιες είναι οι τάσεις για να καθορίσουμε τη μελλοντική πολιτική μας. Λοιπόν, όσον αφορά το τι θα γίνει στο μέλλον, δύο πράγματα θα ήθελα να επισημάνω. Θα αναθεωρήσουμε την οδηγία για τη συνοριακή ε, ε, επιβολή των ε, προστήμων της τροχέας, δηλαδή αν οδηγάς σε κάποια άλλη χώρα θα σε βρίσκει το πρόστιμο. Επίσης θα πρέπει να δούμε τις νέες τάσεις όπως η αυτοματοποίηση θα δούμε επίσης το θέμα του εάν θα πρέπει να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση της αφαίρεσης του διπλώματος και θα πρέπει να δούμε επίσης ε, τις συστάσεις ε, για το ποσοστό αλκοόλ στο αίματος. Υπάρχουν κάποιες συστάσεις ε, τελευταία. Τέλος, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με άλλους τομείς που παρακολουθούμε όπως η ταχύτητα ειδικά σε αστικές περιοχές και οι περισπασμοί των οδηγών, τα κινητά όταν οδηγούμε και Βεβαίω υπάρχει και η πτυχή της ασφάλειας αλλά και ζητήματα όπως η μικροκινητικότητα και τα σχετικά. Ευχαριστώ να τα συζητήσω μαζί σας λίγο σύντομα για την παγκόσμια διάσταση, γιατί μίλησα μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που βεβαίως είναι η βασική ε, δουλειά μου ως συντονιστής. Αλλά επειδή ε, έχουμε ηγετικό ρόλο παγκοσμίω έχουμε την να βοηθήσουμε και άλλους. Ε, τον Φεβρουάριο 19 και 20 έχουμε την πρώτη παγκόσμια διάσκεψη του ΟΗΕ για την οδική ασφάλεια από το 2015 στην Βραζιλία Ελπίζω το σχέδιο δήλωσης, το οποίο είναι διαθέσιμο, να υιοθετηθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο αυτό να υπάρξει ξανά δεσμεύση για παγκόσμιους στόχους. Η Επίτροπος Βαλεάν θα παραστεί, θα μιλήσει στην έναρξη του συνεδρίου, ελπίζω να υπάρξει και εκπροσώπηση των Ευρωβουλευτών και μην ξεχνάμε όταν μιλάμε για τους θανάτους υπολογίζουμε ότι είναι 1,3 εκατομμύρια παγκοσμίω ε, στους δρόμους και θα είναι 40 εκατομμύρια μέχρι το 2050 εάν δεν τα καταφέρουμε και 2050 βεβαίω, υποτίθεται ότι εμείς θέλουμε να φτάσουμε στο 0 εντάξει αν δούμε τις αισθανά ε, θανάτου δεν είναι στο επίπεδο του AIDS ή της φυματίωσης ε, οι δρόμοι είναι πολύ πιο φωνικοί λοιπόν για πρώτη φορά, η δήλωση αυτή για πρώτη φορά σαφή την σχέση μεταξύ οδικής ασφάλειας και βιώσιμων μεταφορών. Είναι εξαιρετική και ελπίζω να τη δείτε. Για να δω τις διάφορες σχέσεις που τονίζουμε. Έχουμε πρώτα απ' όλα το πράσινο deal. Αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να μειωθούν οι εκπομπέ κατά 90% μέχρι το 2050 και να γίνουν τελείω ουδέτερες οι μεταφορές. Λέμε ότι όλες οι μορφές κινητικότητας πρέπει να γίνουν το ίδιο είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Τώρα δεν θέλω να προδικάσω ούτε τη νέα μας στρατηγική, ούτε την επίτροπο που δεν έχει έρθει στην επιτροπή σας, αλλά αναμένω τον ρόλο μου συντονιστή σε αυτό το υπαρξιακό ερώτημα. Παραδείγματο χάρη για κάτι το οποίο μας αφορά η Κομισιόν σκοπεύει να είναι κλιματικά ουδάτερη μέχρι το 2030 και ελπίζω να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο για να το επιτύχουμε αυτό σε σχέση με αυτό αξιολογούμε το πακέτο αστικής κινητικότητας. Προφανώς ε, δεν έχουμε τόσο πολλές αρμοδιότητες ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχει μεγάλη ζήτηση στο τοπικό επίπεδο για ασφαλέστερες ε, μετακινήσεις. Σκεφτείτε την τεράστια συμμετοχή. Χίλιες πόλεις βρίσκονται σε σχετικά σχέδια. Έχουμε εκδώσει κάποιε κατευθυντήριε γραμμές και προσπαθούμε τώρα να φτιάξουμε κάποιου τυποποιημένου δείκτε για να αξιολογήσουν οι πόλει στην πολιτική τους ε, και υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός ε, για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα κινητικότητα ε, την οποία εσείς στηρίξατε και θα έχουμε εδώ στις Βρυξέλλες το τέλος Σεπτεμβρίου την πρώτη σχετική διάσκεψη. πρέπει να σταματήσω γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν ανέφερα για την κινητικότητα υπηρεσία CITS και μια πιθανώς έξυπνη ε, διάσταση στην αστική ε, κινητικότητα. Θα σταματήσω εδώ. Ελπίζω λοιπόν να σας έδωσα να καταλάβετε λίγα πράγματα για τις δραστηριότητές μου και βεβαίως ε, αναμένω και τις δικές σας τις κατευθύνσεις και αν θέλετε ευχαριστώ να ξαναέρθω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μπόλτουιν για την εισήγησή σας που μας δείχνει ότι πρέπει ακόμα να γίνει μεγάλη προσπάθεια και χρειάζεται και βέβαια προσπάθεια και από πλευράς κατορμελών και από πλευράς πόλεων και από πλευράς μας ως ε, νομοθέτες. Έχουμε λοιπόν τώρα δύο λεπτά ανά ομιλητή. Πρώτα απ' όλα η κυρία Τάλερ. Α, όχι η κυρία Τάλερ, θα δώσετε τη σειρά σας στον συνάδελφό σας. Ο κύριος ε, Νομακόφ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Μπόλτον για την εισήγησή σας. Είναι καλό που ξεκινάμε τη φετινή χρονιά με ένα τόσο σημαντικό θέμα που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές. Πέρυσι πρότεινα πιλωτικό πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευτυχώς εγκρίθηκε για τον χειρισμό των ε, απατών στα ταχύμετρα. Ελπίζω αυτό εφαρμόστηκε και ελπίζω πως θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα συντόμως. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε την ανώνυμη ανταλλαγή δεδομένων κάθε ε, ε, ετήσιου συστήματος δοκιμασίας που υποχρεούνται να περνάνε τα οχήματα ώστε να προλαμβάνονται αυτοί οι έμποροι ε, αυτοκινήτων ε, <coughs> που δεν είναι καινούρια και που χρησιμοποιούν διάφορων ειδών απάτες. Ε, θα ήθελα τώρα να πούμε ότι έχοντας υπόψη ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των αυτοκινητιστικών συμβαίνουν λόγω της συμπεριφοράς του οδηγού, ορισμένα οφείλονται στις συνθήκες των δρόμων, αλλά ένα τμήμα οφείλεται στην κατάσταση του ίδιου του αυτοκινήτου. Δυστυχώς υπάρχουν πολλές κοινωνίε σε ολόκληρη την Ευρώπη που δεν μπορούν να αγοράσουν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο και πρέπει να ε, ε, ε, αγοράσουν μεταχειρισμένο. Τι σας λέει η ιδέα για μια πανευρωπαϊκή εγγύηση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου που θα εγγυάται ότι τουλάχιστον κάποια χιλιόμετρα ή κάποια χρονική περίοδος για κάθε πελάτη ιδιοκτήτη μεταχειρισμένου αυτοκινήτου θα έχει έτσι εγγύηση ότι το αυτοκίνητό του δεν θα χαλάσει ή ότι εν πάση περιπτώσει δεν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα ή βλάβη. Επίσης θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι τα μελλοντικά βήματα που προτίθεστε να λάβετε τα επόμενα χρόνια ώστε να εκπαιδεύσετε τους νέους ε, οδηγούς πώς να οδηγούν με μεγαλύτερη ασφάλεια ειδικά σε περίπλοκες καιρικέ συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Δανίελσον έχει το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπόντουιν για την παρουσίασή του. Η οδική ασφάλεια, όπως είπατε, είναι ένα σημαντικό θέμα που μας επηρεάζει όλους, ως επιβάτες, ως εργαζόμενους, ως ποδηλάτες, πεζούς. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τις ε, ε, ενέργειες για να αντιμετωπίσουμε την κατανάλωση αλκοόλ από τους οδηγούς. Θα στηρίζατε ένα όριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους επαγγελματίες οδηγούς. Ένα όριο δηλαδή κατανάλωση αλκοόλ που θα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη, κάτι που δεν συμβαίνει τώρα. Επίσης, θα μπορούσατε να μας πείτε την άποψή σας σε σχέση με το πώς μπορούμε να αυξήσουμε την χρήση των συστημάτων αχινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση ε, κατανάλωσης αλκοόλ από τον οδηγό. Επίσης, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για την υιοθέτηση της οδηγίας για την ασφάλεια των υποδομών. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι όσο το δυνατόν περισσότερα χιλιόμετρα ορίζονται από τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της οδηγίας έτσι ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια στους δρόμους. Σε ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η οδική ασφάλεια είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Όλοι πιστεύω συμφωνούμε. Είδαμε τους αριθμούς, κύριε Μπόλτουιν, και είδαμε ότι αυτή τη στιγμή κατά κάποιο τρόπο η γραμμή είναι ε, επίπεδη, δεν μειώνονται τα ατυχήματα. Θεωρείτε ότι με την αυτόνομη οδήγηση και με την αυτοματοποίηση θα μειωθούν τα ατυχήματα είναι αυτό το κλειδί έτσι ώστε να μειώσουμε το ανθρώπινο σφάλμα. Και πώς διασφαλίζουμε ότι τα αυτόνομα οχήματα επικοινωνούν με σωστό τρόπο. Δηλαδή, όταν εμείς οδηγούμε ένα αυτοκίνητο, βλέπουμε μπροστά μας, αν υπάρχει κάποιος άλλος, μπορούμε να φρενάρουμε. Στις Βρυξέλλες ιδιαίτερα, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, ειδικά για μένα που από τη Γερμανία. Πώς διασφαλίζουμε όμως, πώς θα διασφαλίσουμε μάλλον ότι τα αυτόνομα οχήματα θα επικοινωνούν με σωστό τρόπο. Μας μιλήσατε για το πιλωτικό πρόγραμμα. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες ενδείξεις για τα αποτελέσματα. Παρόλο που θα τα έχετε το Φλεβάρι τα αποτελέσματα τα τελικά, μπορείτε ίσως να μας δώσετε κάποιες ενδείξεις για το τι έχετε βρει μέχρι στιγμής. Ο κύριος Ντάνιλσον μίλησε για το αλκοόλ. Εγώ θα συμπεριλάμβανα σε αυτό και ναρκωτικές ουσίες. Και πράγματι το ζήτημα έχει να κάνει με το ανθρώπινο σφάλμα. Και πώς διασφαλίζουμε επίσης ότι και το ίδιο το όχημα είναι ασφαλές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπόλτουιν για την παρουσίασή του. Είναι καλό το ότι για μια δεκαετία είχαμε καλύτερους αριθμούς, μια βελτίωση, ωστόσο βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει υπάρξει αρκετή πρόοδος. Αναφέρθηκε το ζήτημα των περισπασμών και όταν ε, βλέπουμε ότι πλέον τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν οθόνες όπου μπορούμε να παίξουμε βίντεο από το YouTube και να βλέπουμε και τα μηνύματα στο κινητό μας, θεωρώ ότι αυτό εγείρει ζητήματα σε σχέση με το κατά πόσον όλες αυτές οι συσκευές συμβάλλουν ίσως το πρόβλημα και δεν το επιλύουν. Το ερώτημά μου έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε ε, την πιο ενεργή μετακίνηση, δηλαδή να περπατούν οι άνθρωποι, να χρησιμοποιούν το ποδήλατο, να κάνουν κάτι καλό για την υγεία τους, να καταπολεμούν την παχυσαργία και να κάνουν και ε, κάτι καλό και για την ασφάλεια. Πώς μπορούμε λοιπόν τους πεζούς και τους ποδηλάτες να τους προστατεύσουμε. Υπάρχουν μάλιστα κάποιες πόλεις οι οποίες προωθούν τα αυτοκίνητα και άλλα αυτοκινούμενα οχήματα και όχι την μετακίνηση με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Πώς μπορούμε λοιπόν να προωθήσουμε και πάλι την χρήση του ποδηλάτου ε, και το περπάτημα έτσι ώστε να μπορούμε παράλληλα και τα παιδιά να κυκλοφορούν στους δρόμους χωρίς να φορούν διακριτικά ε, που τα κάνουν να φαίνονται σαν εργάτες και χωρίς να χρειάζεται οι γονείς να τα πηγαίνουν παντού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν κύριε να αναφέρετε το Όσλο. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα όπου αυξάνονται οι ποδηλάτες και οι πεζοί αλλά και προστατεύεται η ασφαλειά τους. Φαντάζομαι η απάντηση έχει να κάνει με το ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερο σχεδιασμό, βελτίωση του δημόσιου χώρου, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τη σκέψη σα γι' αυτό. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά κυρία Ντεσάντου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μπόλντουιν για την ε, πλήρη σας εισήγηση. Ενώ η ασφάλεια στους ε, δρόμους έχει βελτιωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το είπατε πριν από λίγο, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών παραμένει ε, υψηλά. Σε Συμφωνούμε για αυτό το θέμα. Αυτό ε, σημαίνει 25.000 ε, θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 135.000 τραυματίες. Για τη χώρα μου, τη Γαλλία, το 2018 είχαμε 3.400 ε, ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στους, στους δρόμους και 57.000 τραυματίες. Αξιοθρύνητος απολογισμός. Είναι το κόστος όμως αυτό μεγάλο και αφορά και το σύνολο των εργαζομένων πεζωμένο στους δρόμους έχουμε ανταγωνισμό από εργαζόμενου που έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το δίκτυο ερευνητών δημοσιογράφων, το Investigate Europe, ο αριθμός των εγγράφων που επιτρέπει στους εξοκοινοτικούς οδηγού να εργάζονται εντό τη Ένωσης είχε αυξηθεί κατά 286% ανάμεσα στο 2012 και το 2017 και είχε φτάσει στον αριθμό ρεκόρ 108.000. Ε, Μολδαβοί, Λευκορώσοι, ε, Καζακ Καζάκι, ακόμα και ε, τα Ελλαδί ε, ε, ανταγωνίζονται μεταξύ τους και αυτή η παράνομη πρακτική τους αναγκάζει να οδηγούν όσο γίνεται περισσότερο χρονικό διάστημα με τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Γιατί λοιπόν να μην προστατέψουμε τους χρήστες μας από πρακτικές που δεν επιτρέπουμε εμείς στις δικές μας εταιρείες. Η ασφάλεια των δρόμων θα κέρδιζε από κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λεσάντο. Η κυρία Κουντουρά έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, ε, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Baldwin για την παρουσίασή του και να τοποθετηθώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παγκόσμιος ηγέτη στην οδική ασφάλεια. Παρατηρούμε, όπω πολύ σωστά υπόθηκε, μια στασιμότητα στην πρόοδο αφορά τη μείωση των θανάτων από τα τροχαία ατυχήματα τα τελευταία πέντε χρόνια και το 2010 Είδαμε μέχρι το 2013 ότι η μέση ετήσια πρόοδος στη μείωση του αριθμού των θανάτων από τα τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 2,8% και το μεγαλύτερο μέρος ήταν ε, Τη μείωση ανάμεσα στο 11, 12, 13. Από τότε υπάρχει όντω μία στασιμότητα. Δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδο, αλλά υπάρχει και άλλο ένα ανησυχητικό στοιχείο που είναι οι μεγάλες ανισότητες που παρατηρούνται ανάμεσα στα κράτη-μέλη και γνωρίζουμε ότι η οδική ασφάλεια είναι μεν περίπλοκο ζήτημα Απαιτεί δε τη συνεργασία των κρατών μελών, αλλά για να σχεδιάσουμε μια αποδοτική πολιτική θα πρέπει να αναλύσουμε τα κενά των πολιτικών μας μέχρι σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πρώτον πού οφείλεται αυτή η στασιμότητα που παρατηρούμε τα τελευταία πέντε χρόνια και ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες των τόσο διαφορετικών επιδόσεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Τέλος, με βάση αυτά τα συμπεράσματα, ποιο είναι το σχέδιο της Επιτροπής για να μειωθούν αυτές οι ανισότητες ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αρκεί μια γενική στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία, ή μήπω θα έπρεπε η Επιτροπή, αντλώντας στοιχεία από μια συγκριτική ανάλυση, να προχωρήσει και σε συγκεκριμένες συστάσεις στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κουντούρα. Κυρία Τάλερ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπολτουίν για την ε, παρουσίασή σας και για την ε, δουλειά που κάνετε σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Χαίρομαι για το ότι μας δείξατε πάλι το αριθμούς της μείωσης ε, των νεκρών και τραυματιών στους δρόμους και έχετε δει και τώρα αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της ε, στασιμότητας. Ε, δεν μειώνονται πλέον αυτοί οι αριθμοί. Έχω δύο ερωτήσεις. Ε, το πρώτο ερώτημα πηγαίνει προς την κατεύθυνση του κύριου Τιέν που αναφέρθηκε στο θέμα της αυτόματης οδήγησης. Πώς μπορεί η τεχνολογία να αποτελέσει την λύση στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Και η δεύτερη ερώτηση πηγαίνει προς την κατεύθυνση αριθμών και στοιχείων. Έχετε επαρκή στοιχεία από όλα τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να έχουμε μια στέρεη βάση για να γνωρίζουμε γιατί συνέβη ε, το ατύχημα, γιατί υπάρχουν ε, τόσοι νεκροί και τραυματίες, για να έχουμε συγκρίσιμα δεδομένα στα οποία μπορούμε να βασιστούμε για να προγραμματίσουμε τα μελλοντικά βήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Γραφία. Γραφεία. Ευχαριστώ πολύ. Σας, ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας, κύριε Μπάλτουιν. Όπως είπατε σωστά, ο στόχος θα πρέπει να είναι να μειώσουμε τους θανάτους, να φτάσουμε σε μηδενικούς θανάτους στο δρόμο. Ωστόσο, οι αριθμοί παραμένουν τραγικοί. Οι περισπασμοί των οδηγών είναι το βασικό αίτιο των ατυχημάτων. Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Τροχέας, ένα στα τέσσερα ατυχήματα στην Ισπανία προκαλείται από την απόσπαση της προσοχής του οδηγού και την υπερβολική ταχύτητα. Και το βασικότερο στοιχείο που προκαλεί απόσπαση προσοχής είναι το κινητό τηλέφωνο. Αυτό που εγώ θα ήθελα να πω ίσως δεν θα είναι δημοφιλές, αλλά θεωρείτε ότι θα ήταν απαραίτητο να απαγορεύσουμε εντελώς τη χρήση του κινητού τηλεφώνου όταν κάποιος οδηγεί. Έχει υπάρξει ανάγκη να κάνουμε όπως υπάρχει το airplane mode που βάζουμε το κινητό όταν μπαίνουμε στο αεροπλάνο, να υπάρχει ένα, ε, μια αντίστοιχη ρύθμιση και για το αυτοκίνητο που να ενεργοποιείται αυτόματα όταν μπαίνει ο οδηγός μέσα στο αυτοκίνητο. Τι μέτρα θα μπορούσαμε να λάβουμε γι' αυτό. Επίσης, τι μέτρα χρηματοδότησης προβλέπονται στο νέο, στο νέο προϋπολογισμό για την οδική ασφάλεια. Ευχαριστώ. bienvenue à notre euh, député favori, και καλωσορίζω και τον αγαπημένο μας ε, βουλευτή, τον κύριο Βίμ Κάμπο ο οποίος κρύβεται. Καλώς ήρθατε αγαπητέ. Και καλή χρονιά. Έχετε τον λόγο, κύριε Ρικέ, για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπόλουιν. Εγώ έχω κάποιες ε, επιφυλάξεις. Πρώτα απ' όλα, ε, έχουμε μια έκθεση και κάθε φορά βεβαίως ε, μας ε, παρουσιάζεται τις μειώσεις θα πρέπει να μας πλέτε και τον αριθμό χιλιόμετρων που διανύονται γιατί τότε η πτώση είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή σε σχέση με τα χιλιόμετρα τα οποία διανύονται. Δεύτερον, δεν υπάρχει επίσης ε, η σχέση με την αιτία του ατυχήματος, ε, οι οποίες αιτίε αλλάζουν. Δηλαδή, αν είχαμε αυτή την πτώση πριν από 10-15 χρόνια, αυτό οφείλεται κατ' ουσίαν στις ζώνες ασφαλείας που μείωσαν τους ανάτους στο μισό κτλ. Μετά. Μετά είχαμε την εισαγωγή του κινητού τηλεφώνου. Έχουμε μια νέα αιτία των ατυχημάτων. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιος συσχετισμός από πλευρά σας ε, μεταξύ της προόδου και των νέων παραγόντων βεβαίως. Εντάξει, έχουμε και τις νέες τεχνολογικές προόδους που φρενάρουν τα αυτοκίνητα μόνο τους, έχουν την κάμερα οπισθοπορίας και τα σχετικά. Ε, λοιπόν, δεν υπάρχει ερμηνεία άρα λοιπόν σε αυτά τα οποία μας λέτε και δεν ισχύουν. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να κάνουμε την ίδια συζήτηση, δηλαδή προτάσεις όσο που αφορούν τη συμπεριφορά του οδηγού, συστάσεις, ίσως θα ζητήσουμε και θα επιβάλλουμε να οδηγούν 40 ε, την ώρα στις ε, ε, στις εθνικές οδούς και με 10 μέσα στις πόλεις. Σωστά μιλήσατε και για την κατάσταση το στόλου των οχημάτων. Υπάρχει μια διαφορά στην ισορροπία ανάμεσα στο, στην ε, Ανατολή και τη Δύση, δηλαδή δεν είναι πιο ανόητη η οδηγία, ας πούμε, στη Βουλγαρία, η πιο έξυπνη, η Νορβηγή οδηγεί. Ε, και έπειτα, οι ευάλωτοι χρήστες ε, πάντοτε μας ενδιαφέρουν μόνο ως θύματα ή μήπως και ως θύτες και οι υπεύθυνου για τη δική τους ατυχία. Γιατί, εντάξει, μπορούμε να μιλάμε για αυτούς που οδηγούν σαν τρελή, αλλά και η συμπεριφορά των ευάλωτων χρηστών και αυτή είναι πολύ ε, επικίνδυνη. Και βεβαίω, και αυτό θα είναι η τελευταία μου λέξη για να κλείσω, είναι ότι η παρουσίαση των ειδών όπως γίνεται είναι τελείω λάθο. και μάλιστα καταλήγει σε προτάσει, οι οποίε είναι άσκοπες ε, και ατυχεί. Και εδώ θα έλεγα ότι έτσι δεν θα πρέπει να απαλλάξουμε τα κράτη-μέλη από το να εξετάσουν από τους σύνεγγυ ε, την νομοθεσία που φοβά τι υποδομέ, την ποιότητα των οχημάτων και τον έλεγχο αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρικέ. Κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση πολύ ενδιαφέρουσα για τη Γερμανία, γι' αυτό θα συνεχίσω στα γερμανικά. Υπάρχει αυτή η κατάσταση την οποία αναφέρατε που είναι αμοιβαίως υποφελής ε, ε, μεταξύ ασφάλειας και νέων τεχνολογιών. Ε, η ερώτησή μου είναι η εξής. Έχετε υπόψη ε, το ότι έχουμε ένα μοσαϊκό ορίον ταχύτητας πανευρωπαϊκό το οποίο είναι αντιπαραγωγικό. Κάποιες πόλεις θέλουν να προχωρήσουν πιο μπροστά, να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για τους πολίτες αλλά δεν μπορούν γιατί ε, διαφέρουν οι εθνικές νομοθεσίες. Και σκέφτομαι και τον οδηγό ο οποίος ε, παντού ανά την Ευρώπη αντιμετωπίζει διαφορετικά όρια και αυτό είναι μια δυσκολία. Θα μπορούσε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει μια σύσταση λογική βεβαίως ε, για την ασφάλεια των παιδιών ε, και βεβαίως για την κλιματική αλλαγή. Και το τελευταίο ερώτημα που σχετίζεται με αυτό θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει και μια πτυχή του Green Deal. Να πείτε δηλαδή εδώ πέρα θα φροντίσουμε και την οδική ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή. Σας ευχαριστώ κύριε Φλεγκό, έχετε τον λόγο. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς ε, πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ακούσουμε πολύ προσεκτικά τα όσα λέγονται. Εν η ώρα τα αυτόνομα αυτοκίνητα να τα πάρουμε πιο σοβαρά υπόψη και να τα εισάγουμε στις μεταφορές. Έχουν γίνει μελέτες που να μετρούν την ασφάλεια έτσι ώστε επί τη βάση αυτών των στοιχείων να μπορούμε να ε, εξετάσουμε και νομοθετικές λύσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Ολιβιέ έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλήσαμε για, γενικά για οδική ασφάλεια και είναι όλα αυτά πολύ ενδιαφέροντα, αλλά εγώ θα ήθελα να σκεφτούμε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο, δηλαδή την ασφάλεια των μοτοσυκλετιστών. Και θα είμαι πολύ συγκεκριμένο, γιατί το θέμα τη ασφάλεια των μοτοσυκλετιστών είναι πιο ιδιαίτερη, αφορά την ισορροπία του και όσα μπορούν να του προστατεύσουν. Πρώτο προβληματισμό αφορά τι υποδομέ, βέβαια μιλήσαμε γι' αυτό και για του μοτοσυκλετιστέ είναι αρκετά πρακτικό όσον αφορά, α πούμε, τι ε, γούβε που σχηματίζονται συνέχεια. Έπειτα, προσαρμογή των ε, διαφόρων ε, οδικών βοηθημάτων, όπως ας πούμε οι πάσαλοι που δεν, δεν τοποθετούνται σωστά και έπειτα ακόμα και οι, οι βαφές με τις οποίες ε, γίνονται τα διάφορα σήματα πάνω στην επιφάνεια της ασφάλτου είναι ιδιαίτερα ολιστηρές για τους μοτοσυκλετεστές. Ε, και ένα σωρό άλλα εξοπλισμοί ατομική ασφάλειας, ε, δηλαδή κράνος, γάντια, μπότες, ε, ειδικά μπουφάν με airbag, είναι πολύ δαπανηρή εξοπλισμοί, ακριβή εξοπλισμοί και γι' αυτό ίσως θα έπρεπε να μειωθεί η σχετική φορολογία τους. Τελευταία παρατήρηση που δεν αφορά τους μοτοσυκλετιστές μόνο, αλλά περισσότερο αφορά την κατάρτιση αυτών και των οδηγών αυτοκινήτων για την ε, συγκατοίκηση με τους μοτοσυκλετιστές. Πολύ συγκεκριμένο θέμα βλέπετε. Εγώ δεν είμαι ο πιο υπέρ ε, νέων ε, νομοθετημάτων, αλλά στο αυτό το θέμα πιστεύω πως χρειάζονται νέες νομοθεσίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Γραπίνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, από την δική σας παρουσίαση δεν φαίνεται να υπάρχει ταξινόμηση των ατυχημάτων ανάλογα με το αίτιο, δηλαδή αν είναι υποδομές, χρήση αλκοόλ, χρήση ναρκωτικών και ούτω καθεξής. Αν δεν έχουμε μια τέτοια ταξινόμηση δεν μπορούμε να λάβουμε άμεσα μέτρα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα αίτια αυτά. Αν ένα ατύχημα γίνεται λόγω χρήσης ε, ναρκωτικών μπορούμε να προβλέψουμε εναρμονισμένη νομοθεσία και απαγόρευση της χρήσης των ναρκωτικών. Εάν οφείλεται στην ε, ε, μη χρήση της ε, ζώνης ασφαλείας είναι άλλο ζήτημα. Χρειάζεται λοιπόν συγκεκριμένη νέα νομοθεσία που να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Για παράδειγμα, στη χώρα μου αν έχουμε κατόφλι μηδέν, μηδενικής ανοχής χρήσης αλκοόλ, κατανάλωσης αλκοόλ, σε άλλη χώρα μπορεί να είναι διαφορετική η νομοθεσία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν μπορούμε σε μια ενιαία χώρα να έχουμε τέτοιες διαφορές σε αυτό το τομέα, γιατί δεν είναι θετικό αυτό. Πέρα τώρα από τους ε, μοτοσυκλατιστές ή τους ποδηλάτες υπάρχουν και εκείνα τα πατίνια. Δεν χρειάζεται άδεια οδήγηση για τα πατίνια, αλλά ε, μιλάμε για την οικολογική πτυχή της χρήσης τους, αλλά ξέρουμε πόσα ατυχήματα <laughs> προκαλούν τα πατίνια. Είδαμε στα γραφήματά σας ε, τα στοιχεία μέχρι το 17. Πιστεύω όμως ότι όλοι μαζί πρέπει να προβληματιστούμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να ε, φτιάξουμε συγκεκριμένα μέτρα γιατί διαφορετικά μιλάμε για να μιλάμε. Τα νούμερα που μας δείξατε δεν ξέρω καν από πού προέρχονται. Μάλιστα, η κυρία Τάξη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε και στον κύριο Βίμ Φαντεκάμπ. Συμφωνώ λοιπόν, κύριε Μπόλτουιν. Όλοι αυτοί οι αριθμοί είναι πολύ σημαντικοί. Αν συνέβαινε στον τομέα των αερομετωφορών θα είχαμε μια κρίση στην Ευρώπη. Έχουμε ε, έναν οργανισμό για την ασφάλεια στη θάλασσα και για την ασφάλεια στις αερομεταφορές, αλλά όχι έναν οργανισμό για την οδική ασφάλεια. Πριν από κάποιο διάστημα βρέθηκα στις διαπραγματεύσεις για τους χρόνους οδήγησης και ξεκούρασης και διαπίστωσα ότι ένα βασικό πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχουμε τους σχετικούς κανόνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη και το πώς εφαρμόζουν την νομοθεσία. Αν εγώ λοιπόν ήμουν επίτροπος, θα δημιουργούσα μια υπηρεσία οδικής ασφάλειας. Τι πιστεύετε εσείς γι' αυτό? Ευχαριστώ, κύριε Λούτχεν. Ναι, σωστά το είπα το όνομά σας. Ναι, ναι. Είμαι πολύ ευτυχής που το είπατε σωστά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον κύριο Μπόλουιν για την παρουσίαση. Ωστόσο, Δυστυχώς χρειάζομαι ε, να πω και εγώ κάποια πράγματα όπως και ο κύριος Ρικέ, παρότι δεν είμαι εδώ, εδώ και 10 χρόνια. Βέβαια τα νούμερα δεν σχετίζονται με αριθμό χιλιόμετρων που έχουν διανυθεί, οπότε μπορεί ο καθένας να δώσει ό,τι ερμηνεία θέλει. Επίσης, για τα αίτια το είπαν και άλλοι παρεμβαίνοντες, ποια είναι τα αίτια αναχώρα και μέσα σε μια χώρα μπορεί και εκεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις από τη μια περιφέρεια στην άλλη, ας πούμε, ε, ε, ανάμεσα στις περιοχές της υπαίθρου ή τις αστικές περιοχές. Και αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως, δεν ξέρω αν αυτό είναι δυνατόν, ίσως αν δημιουργηθεί μια, ένας οργανισμός για την οδική ασφάλεια να το καταφέρουμε, αλλά να είχαμε ας πούμε συστάσεις ανακάτως ένα μέλος, ώστε να πούμε να, αυτές είναι οι προτεραιότητες όσον αφορά την οδική ασφάλεια, ώστε αυτή η τελμάτωση που είναι και όπως είπα εντό εισαγωγικών γιατί πρέπει να δούμε πόσα χιλιόμετρα, σε πόσα χιλιόμετρα σημαίνονται αυτά τα ατυχήματα. Να μπορεί λοιπόν το κάθε κράτος μέλος να μπορεί να μειώσει δραστικά τον αριθμό θυμάτων από τα αυτοκινητιστικά στη χώρα του, γιατί οι διαφορές είναι τεράστιες ε, όσον αφορά το κατανάλωση αλκοόλ, ναρκωτικών, τον ε, διαφορά ανάμεσα στις υποδομές, ε, το είδος των αυτοκινητών που χρησιμοποιούνται, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και πάλι θα έπρεπε να διασταυρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε συστάσεις, ώστε πραγματικά να ληφθούν μέτρα από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν, αν και εν μέρει τα γνωρίζουν, να ξέρουν ποια θα είναι τα πιο αποτελεσματικά μέτρα που θα μπορούσαν να λάβουν, ανάλογα με την πραγματικότητα που ισχύει και κάτι τέτοιο θα ήταν χρήσιμο αν θέλουμε πραγματικά να προάγουμε την οδική ασφάλεια. Χρειάζεται λοιπόν παρακολούθηση και να μπορούμε κάθε κράτος μέλος να μπορεί να παρακολουθήσει βήμα-βήμα και εθνικοί περιφερειακοί βουλευτές να μπορούν να παρακολουθούν τα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με τις συστάσεις που θα έχει ε, υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αρμό έχει τώρα το λόγο. Εγώ δεν θα επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν, αλλά αν δούμε τα πόσα χιλιόμετρα διανύονται σε κάθε χώρα, υπάρχουν ε, διαφορές 1 ε, μέχρι 10. Έγινε λόγος για τελμάτωση, αλλά υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη όπου ο αριθμός των θανάτων αυξάνεται. Δηλαδή είμαστε τυχεροί ακόμα και αν ορισμένε χώρες ε, έχουν σταθεροποιηθεί, κάποιες άλλες όμως αυξάνονται. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν μεγάλες ε, διαφοροποιήσεις και αυτό για διαφορετικές αιτίε. Ας πούμε στη Ρουμανία δεν επιτρέπεται να οδηγεί κανείς όταν έχει αλκοόλ στο αίμα του, δηλαδή υπάρχει μηδενική ανοχή στην κατανάλωση αλκοόλ. Δηλαδή πρέπει να μπορούμε να δούμε σε επίπεδο ένωσης Key Performance Indicators, δηλαδή δείκτες ε, ε, επιδόσεων και να μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή την πείρα της Δύσης στις χώρες της Ανατολής, γιατί στις χώρες μας αυξάνεται η χρήση των αυτοκινήτων. Οι άνθρωποι δεν είχαν αυτοκίνητα, πολύ πρόσφατα απέκτησαν Οπότε πρέπει να υπάρχει ένα είδος μεταφοράς τεχνογνωσίας για να λύσουμε τα προβλήματα περιφέρεια προς περιφόρεια. Μια σχέση 1 προς 10 είναι τεράστιο. Δεν μπορούμε δηλαδή να βγάζουμε ένα μέσο όρο και να λέμε ότι ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Ε, στις χώρες όπου το πρόβλημα είναι πιο έντονο θα πρέπει να ασκηθούν συγκεκριμένες πολιτικές και να βοηθηθούν οι κυβερνήσεις τους. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κυρία Αρμό. Κύριε Ντελή. Το θέμα αυτό ήδη αναφέρθηκε από την συνάδελφο δηλαδή τις εναλλακτικές μορφές μετακίνησης της πόλης, είτε πρόκειται για segway, πατίνια και άλλα οχήματα. Η λογική είναι πολύ απλή, μειώνονται οι εκπομπές, μειώνεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Παρόλα αυτά όμως, εγείρουν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια όλων των χρηστών του δρόμου, όχι μόνο για τους ίδιους. Υπήρξε το ζήτημα της ευαλωτότητας και το κατά πόσον αυτοί οι χρήστες είναι ευάλωτοι. Ίσως θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιες ε, κατευθυντήριες γραμμές, κάποια ελάχιστα πρότυπα για τις πόλεις, για το πώς μπορούν δηλαδή οι πόλεις να οργανώσουν τέτοιου είδους μετακινήσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ανταγωνισμός των τρόπων μεταφοράς μέσα στις πόλεις. Αναφέρετε επίσης στην παρουσίασή σας την διασυνοριακή εφαρμογή των παραβιάσεων της τροχέας το δοκίμασα και λειτουργεί. Δηλαδή, το έχω δει στην πράξη. Τι θα κάνετε όμως εσείς, έτσι ώστε να λειτουργεί περισσότερο αυτό το θέμα. Αυτό ο τομέας είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεφύγει κανείς από μια τροχιά ε, παράβαση. Οπότε, ποιε είναι οι σκέψει για το πώ μπορούμε να αυξήσουμε την εφαρμογή αυτή τη νομοθεσία. Σα ευχαριστώ πολύ και είχα και εγώ μια τελευταία ερώτηση. Πολλά ερωτήματα έχουν υποβληθεί, ναι. Εγώ πιστεύω ότι εξαρτάται ο αριθμός νεκρών στους δρόμους μας από πολλές παραμέτρους, αλλά θα ήθελα να επανέλθω σε μια παράμετρο βασική κατά τη γνώμη μου, που είναι η ταχύτητα. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας ε, στη ατυχήματα. Έχουμε νούμερα λοιπόν για αυτό το παράγοντα της ταχύτητας. Επίσης, πολλοί συνάδελφοι είπαν, μίλησαν για το πότε θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι κατεξοδότητες πράξεις για τα, αυτό, την, αυτόνομη οδήγηση και θα, αύριο μεθαύριο θα έχουμε δείκτες και για την ε, ε, ταχύτητα και έπειτα. Βλέπω αυτό που, αυτό που συμβαίνουν και που μου δημιουργούν πολλά ερωτήματα. Δεν θα σας διοικηθώ την ιστορία της ζωής μου, αλλά υπάρχει κάτι όχι, όχι, δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό, αλλά συμβαίνει κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Στις πόλεις είδαμε να φτάνουν τα SUV, αυτά τα Sport Utility Vehicles. Όταν βλέπω λοιπόν τις εφημερίδες, κάθε φορά που βλέπω να γίνεται ένα τύχημα, το τελευταίο που είδα ήταν στο Βερολίνο, υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο βάρος ενός οχήματος και την οδική ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω από ένα τέτοιο όχημα και, και εν γέννη πρόκειται για τους πιο ευάλωτους. Και ακόμα και αν ε, γίνει ατύχημα ανάμεσα στο SUV και ένα άλλο αυτοκίνητο, ε, συνήθως το SUV είναι αυτό που προκαλεί περισσότερες ζημιές ε, γύρω του, εν πάση περιπτώσει, μόνο και μόνο λόγω του βάρους του εσείς έχετε μια γνώμη γι' αυτό, γιατί όταν έχουμε τόσο βαριά αυτοκίνητα αύριο μεθαύριο δεν σημαίνει αυτό ακόμη περισσότερους κινδύνους στους δρόμους. Και ξέρω πως έχει γίνει και μια πρόσφατη μελέτη από τον Οργανισμό για την Οδική Ασφάλεια της Βαλονίας που κάπως το είχε, είχε επικεντρώσει σε αυτό το θέμα. Δεν πιστεύετε εσείς λοιπόν ότι το βάρος των αυτοκινήτων αυτών που είναι, θα είναι ένας από τους μεγάλους εχθρούς ε, της οδικής ασφάλειας στο μέλλον. Υπάρχουν μήπως άλλες ερωτήσεις. Όχι. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, αλλά εσείς ε, πρέπει να μας δώσετε πολλές απαντήσεις. Κύριε έχετε το λόγο. Πόσο χρόνο μου δίνετε. Άντε, 12 λεπτά γιατί όπως είπατε, οι ερωτήσει ήταν φανταστικές. Μια εβδομάδα θα μπορούσαμε να περάσουμε συζητώντας τις. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα πρέπει να έρχεστε σε επαφή μαζί μου, να με ε, τσιγκλίζετε και να μου θέτετε αυτές τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Για την απάτη. Έχουμε νέους κανόνες που άρχισαν να ισχύουν για το 2000, από το 2018 και έχετε δίκιο, δίκιο ότι η ανταλλαγή ε, στοιχείων είναι αυτή που περιορίζει την ε, δυνατότητα απάτησης στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα όσον αφορά τις ε, απάτες στους χιλιομετρητές γίνονται πολλές ε, προσπάθειες. Θα πρέπει να εκφράσω κάποιους δισταγμούς για την ιδέα του να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ο αστυνόμος ε, που θα επιβλέπει όλους τους πολιτές ε, μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Για την εγγύηση δε, που είπατε για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι καλή ιδέα, αλλά δεν, στην δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ένωσης. Τώρα, ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης αποφασίζουν τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με την οδηγία για τις άδειες οδήγησης, ε, όλο είναι και περισσότερες εκκλήσεις γίνονται όσον αφορά την εναρμόνιση των μαθημάτων για την άδεια οδήγησης, γιατί όταν περνά τα σύνορα η οδηγοί υπάρχουν κάποια, ε, κάποια προβλήματα και πρέπει να υπάρχουν κανόνες διασυνοριακοί ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια κατάρτιση για τους επαγγελματίες οδηγούς και το αλκοόλ. Α, ναι, συγγνώμη, ξεχνάω που κάθεστε κάθε φορά. Έχω σημειώσει τα ονόματά σας, κύριε Ντάνιελσον. Η σύσταση είναι 0,2 όριο για τους νέους οδηγούς και για τους επαγγελματίες οδηγούς, αφορά την κατανάλωση αλκοόλ. Άλλε ερωτήσει τώρα που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ. Ναι, θα τα αναθεωρήσουμε αυτά τα όρια το μέλλον. Τώρα όλα τα κρατη με μια εξαίρεση που είναι η χώρα μου, το συστηνόμενο επίπεδο για τη συνολική, ε, το συνολικό όριο κατανάλωση αλκοόλ είναι το 0,5. Αλλά πολλές χώρες πάνε στο 0. Ή, εν πάση περιπτώσει, 0,2 είναι σχεδόν 0 όσον αφορά την ανοχή στο αλκοόλ. Ενδιαφέρουσε ιδέε για το αν και πώς θα προχωρήσουμε περισσότερο αυτό, όμω, όπω και η ταχύτητα είναι και θέμα και αρμοδιότητα των κρατών μελών γιατί ο κώδικας κυκλοφορίας είναι θέμα κράτους μέλους. Εμείς κάνουμε προτάσεις, κάνουμε συστάσεις προς τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει να κάνει και με την επιβολή, με την ανείχνευση, το πώς θα μπορέσουμε να πιάσουμε τους παραβάτες. Είμαι κατά λοιπόν, θέμα... δεν είμαι κατά μάλλον ως θέμα αρχής, το εξετάζουμε. Αλλά σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να δεσμευτώ ότι εμεί θα προχωρήσουμε περισσότερο όσον αφορά τα όρια κατανάλωσης αλκοόλ για του επαγγελματίε οδηγού ή το ευρύτερο κοινό. Τώρα, για τις υποδομές. Σας ευχαριστώ καταρχάς για όλη τη δουλειά που έχετε κάνει. Έχουμε πολύ ισχυρότερη οδηγία. Πώς εξασφαλίζουμε μέγιστο αντίκτυπο. Μία από τις συμβιβαστικές ήταν ότι θέλαμε να καλύπτονται όλες οι εθνικές οδοί και επιτρέψαμε τελευταία συμβιβαστική τα κάτι μέλη να μπορούν να ζητήσουν εξαιρέσει για κάποιους εθνικές οδούς. Το θέμα είναι ότι να είναι πραγματικά και δίκαια, πραγματικές και δίκαιες αυτές οι εξαιρέσεις, αλλά για να έρθουμε στους δρόμους των TEN-T ε, θα βάλουμε εκεί και τους αυτοκινητόδρομους και εκεί θα έχουμε σημαντική διαφορά φορά από ό,τι λένε τα στοιχεία. Και κάτι άλλο, για πρώτη φορά επίσης θα απαιτήσουμε από τα κατημέλη να λάβουν υπόψη τις ανάγκες των ευάλωτων χρηστών των δρόμων στο σχεδιασμό των οδικών τους υποδομών. Κύριε Έτγεν, για τα αυτόματα οχήματα, τεράστια ερωτήματα για το ποιο θα είναι τα αποτελέσματα. πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι αυτές οι εξελίξεις θα αυξάνονται θα ε, περάσει πολύ καιρό μέχρι ότου να μπορούμε να μιλάμε για κυρίω αυτοματοποιημένα οχήματα, δηλαδή επίπεδο 4, που βασικά ο, το αυτοκίνητο κάνει όλη τη δουλειά. Θα περάσουν δεκαετίε δεδομένου του χρόνου ζωής των οχημάτων, ε, μέχρι ότου να λειτουργήσουν όλα αυτά. Τα επόμενα 20-30 χρόνια λοιπόν θα έχουμε αυτοκίνητα με διάφορα επίπεδα αυτοματοποίησης που θα συνεπάρχουν. Και αυτό που είπατε είναι πολύ έγκυρο. Υπάρχει ένας βελγικός τρόπος ε, ε σημάτων ε, στα, στα σταυροδρόμια και η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων παίζει ρόλο. Και στο μέλλον θα έχουμε επικοινωνία μεταξύ ανθρώπου και μηχανήματος και ανάμεσα σε μηχανές. Πολύ περίπλοκο ε, ζήτημα. Πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι λοιπόν σε όλα αυτά. Αυτό είναι το αντικείμενο της μελάτη και ευχαριστώ και πάλι το Κοινοβούλιο που το χρηματοδότησε. Δεν μπορώ να σα πω στοιχεία γιατί δεν έχω δει ακόμα τη μελέτη και τα πορίσματά τη. Οπότε θα το συζητήσουμε βεβαίως με μεγάλο ενδιαφέρον μόλις θα εκδοθεί η εν λόγω μελέτη. Κάτι ακόμα που ήθελα να πω για την αυτοματοποίηση εν γέννη είναι ότι συχνά λέγεται ότι ότι είναι η ίστατη μαγική λύση στην ασφάλεια, την οδική ασφάλεια, γιατί βγάζουμε τον άνθρωπο από την εξίσωση. Και όπως είπαμε συχνά, το 90% των ατυχημάτων οφείλεται σε το ανθρώπινο σφάλμα. Εγώ όμως ε, λέω και σας ειδοποιώ ότι ναι, τα σφάλματα είναι λάθος, αλλά μόνο στους δρόμους το σφάλμα ενός ε, οδηγού μπορεί να σε σκοτώσει. Ας πούμε, αν μου πέσουν τα κλειδιά, είναι ανθρώπινο σφάλμα, αλλά δεν θα με σκοτώσει. Ο θάνατος είναι η ίστατη ποινή για ένα σφάλμα που μπορεί να κάνεις. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε τους ανθρώπους, κατά, να, να, τους μάθουμε να, να δρουν ενάντια στα ίδια τους τα σφάλματα. Όμως βραχυπρόθεσμα οι άνθρωποι είναι καλοί στα αυτά που κάνουν και ακόμα και τα καλύτερα μηχανήματα μόλις αρχίζουν κάπως να μοιάζουν με οδηγή. Και όχι καλύτερη οδηγή. Λοιπόν, ας μην βιαστούμε, ας μην βιαστούμε για να χρησιμοποιήσουμε την αυτομετωπίση ως ίστατη λύση για την οδική ασφάλεια. Υπάρχουν πτυχέ τη αυτοματοποίησης που μπορούμε και θα έπρεπε να βάλουμε στα συστήματα οδήγησής μας και το κάναμε. Και πάλι χάρη σε εσά το Κοινοβούλιο με τον νέο γενικό ε, κανονισμό για την ε, αυτοματοποίηση έχουμε βάλει πράγματα όπως α πούμε αυτόματο φρενάρισμα, ε, που θα βοηθήσει στη μεγαλύτερη ασφάλεια των ανθρώπων εντός και εκτός των αυτοκινήτων. Κύριε Κοφέ, ευχαριστώ πολύ για τι παρατηρήσει σα. Είναι πραγματικά ενοχλητικό να βλέπει κανεί ε, την τελμάτωση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ε, δεν μπορούμε, βλέπουμε αύξηση των θανάτων που οφείλεται σε αφηρημένους οδηγούς. Η απόσπαση, η αφηρημάδα μπορεί να προέρχεται από διάφορα πράγματα, από τα συστήματα του αυτοκίνητου, ας πούμε, ε, τηλέφωνα, διαφημίσεις που εκτός, από, εκτός του αυτοκίνητου και πρέπει να έχουμε μια γενική εικόνα. Αν ε, ε, υπάρχει ένας ρόλος που μπορούν να παίξουν οι τεχνολογίε, είναι να εμποδίσουν αυτά τα ατυχήματα και τις, την απόσπαση της προσοχής. Συμφωνώ μαζί σας για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε την δραστήρια μετακίνηση. Εκεί συνδυάζεται η ασφάλεια, η οδική και η βιώσιμη κινητικότητα. Πώς γίνεται αυτό μέσω της διαχείρισης της ταχύτητας. Θα πω περισσότερα απαντώντας στην παρατήρηση της κυρία Ντέλη. Τα, τα στοιχεία ξεκινούν. Όταν σε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο σαν πεζό, ενώ το αυτοκίνητο τρέχει με 30 χιλιόμετρα την ώρα, έχεις 90% πιθανότητες να επιβιώσεις. Ενώ αν σε χτυπήσει τρέχοντας με 60 χιλιόμετρα, οι πιθανότητες να επιζήσεις πέφτουν στο 10%. Οπότε πιστεύω πως δεν χρειάζεται πολύ να ψάξουμε ακόμα, ώστε να πούμε ότι ναι, πρέπει να ισχύει η ταχύτητα των 30 χιλιόμετρων την ώρα μέσα στις αστικές, στα αστικά κέντρα και για πρώτη φορά η δήλωση της Στοκχόλμη μιλά γι' αυτό. Η ταχύτητα είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν βελτιώσεις των υποδομών βεβαίω. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι σχετικά ε, φτηνά ε, και βοηθούν στην ασφάλεια. Και μιλήσατε και για το παράδοξο σχήμα. Ε, σαν νέος γονιός μπορεί να αποφασίσεις σε μια πόλη σαν τις Βρυξέλλες να πηγαίνεις τα παιδιά σου στο σχολείο γιατί ακριβώς ανησυχείς για την ασφάλειά τους από τα αυτοκίνητα. Και άρα είσαι και σε άλλο ένα αυτοκίνητα στο δρόμο και άρα όλο ένα και δυσκολότερο γίνεται για τους γονείς που θέλουν να περπατήσουν αφήσουν τα παιδιά του στο σχολείο ή να πάνε με το ποδήλατο. Θα πρέπει, όπω είπατε, να, να, να, να θεωρείται πλέον φυσιολογική μετακίνηση με τα πόδια με το ποδήλατο. Αναφερθήκατε στο Όσλο. Α μιλήσω για τι Βρυξέλλε και θέλω πραγματικά να συμβάλλω και, και να επενέσω τη δουλειά που γίνεται στην περιφέρεια των Βρυξελών με τι καλέ κινήσει που κάνουν για βελτίωση τη οδική ασφάλεια και πραγματικά είμαι πανευτυχή που θα επιβληθεί όριο 30 χιλιόμετρων την ώρα μέσα στην ε, ε, ε αστική περιοχή των Βρυξελών με λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα στον περιφερειακό. Αυτό σημαίνει τοπική δράση, βελτίωση της οδικής ασφάλειας τοπικά και βιώσιμες δυνατότητες μετακίνησης. Ναι, υπάρχουν τώρα στοιχεία τα οποία εξακολουθούν να είναι πολύ ψηλά. Είναι πολύ κρίμα και σας ευχαριστώ που το αναφέρατε η αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων που σχετίζονται με τους οδηγούς των, με, τους, με τους εργαζόμενους στους δρόμους όπως οι οδηγοί από τη Μολδαβία, από τις Φιλιππίνες που εργάζονται στους δρόμους μας. Συμφωνώ απολύτω μαζί σας ότι είναι πρόβλημα, είναι όμως εκτός της δικής μου δικαιοδοσίας για το, την προέλευση των ανθρώπων. Εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ, ε, ε, με προβληματίζει η ασφάλεια των εργαζομένων στους δρόμους και αυτών ας πούμε, που διορθώνουν τους δρόμους, που επισκευάζουν τους δρόμους. Πολλοί κόσμος περνά δίπλα τους με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ξέρω πως δεν με ρωτήσατε για αυτό το πράγμα, αλλά ελπίζω πως θα μπορέσουμε να το δούμε και αυτό σύντομα, γιατί είναι γι' αυτό πολύ ανησυχητικό. Κύριε Κοντούρου, τελμάτωση. Κυρία Κουντουρά, συγγνώμη, τελμάτωση. Ε, ποιοι είναι οι παράγοντε, Πολλοί λένε πώ ξέρουν τι προκαλεί τα ατυχήματα και τα θύματα αυτών. Πολύ συχνά λέει ο κόσμος, να ξέρω ακριβώ τι ισχύει. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι πρόκειται για ένα κοκτέιλ παραγόντων και επανέρχομαι στο ασφαλές σύστημα που έλεγα πριν. Σε οποιαδήποτε ατύχημα, ένα σφάλμα σχεδόν αναπόφευκτα έχει γίνει. 90% ε, υπάρχει σφάλμα, αλλά το σφάλμα δεν είναι πάντα το αίτιο του θανάτου. Ας πούμε, αν οι υποδομές είναι σωστές, αν η ταχύτητα είναι χαμηλή, εάν ο προστατευτικός εξοπλισμός χρησιμοποιηθεί, τότε μπορεί να, δεν είναι απαραίτητο ότι θα υπάρξει σοβαρός τραυματισμός ή ε, θάνατος και είναι πολύ σωστό που επιστήνετε την προσοχή, σας, στην, την προσοχή μας στις διαφορές που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ένωση και πάλι με τη στήριξη των εταίρων έχουμε ξεκινήσει με το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας και να θυμίσω και την Έλληνα Townsend που είναι σημαντικός εταίρος μας, το Συμβούλιο δηλαδή Οδικής Ασφάλειας, δουλεύουμε με έξι χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Λιθουανία όχι για να κατονομάσουμε ή να καταδείξουμε, αλλά για να συνεργαστούμε, να μειωθούν ε, τα φρικτά, ε, ε, οι φρικτοί θάνατοι στους δρόμους που εξακολουθούν να υπάρχουν. Είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Δουλεύουμε, ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Ναι, ανάμεσα στην Δυτική και την Ανατολική και Νότια Ευρώπη, ώστε να δουλέψουμε και όχι μόνο προς μία κατεύθυνση μόνο. Νομίζω πως η Βουλγαρία έχει μια ιδιαίτερα ε, καλή δουλειά που κάνεις με την ελάφρυνση των ε, επιπτώσεων των ατυχημάτων. Κυρία Τάλερ. Τα στοιχεία, ναι, ε, υπάρχουν εκεί όπου υπάρχουν, αλλά η τεχνολογία πώς μπορεί να αποτελέσει ένα παράγοντα σημαντικό Από το 2022 λοιπόν όλα τα οχήματα που είναι νέα μοντέλα θα πρέπει να περιέχουν κάποια από τα στοιχεία ασφάλεια που προβλέπονται από τον Κανονισμό Γενική Ασφάλεια και όλα τα αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά μέχρι το 2024. Η τεχνολογία λοιπόν μπορεί να μας βοηθήσει πολύ αν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά έτσι ώστε να αυξήσουμε την οδική ασφάλεια. Σε ό,τι αφορά την κατανόηση των λόγων για τους οποίους τα ατυχήματα σκοτώνουν τους ανθρώπους. Αυτό κάνουν τα στοιχεία των ε, δικτών επίδοσης που ανέφερα προηγουμένως. Το 2020 λοιπόν θα αρχίσουμε ε, να εφαρμόζουμε αυτούς τους δείκτες και θα ενημερώσω την Κομισιόν ε, σχετικά. Επιπλέον θα πρέπει να μάθουμε και από το, κάθε οδικό ατύχημα. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, αλλά και στις Ηνωμένε Πολιτείε γίνεται μια σχετική προσπάθεια, δηλαδή προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία από κάθε οδικό ε, ατύχημα. Δηλαδή, μέσα από το αυτοκίνητο να δούμε πόσο γρήγορα πήγαινε, ποια ήταν η κατάσταση του οδοστρώματος, ε, κατά πόσο ο οδηγό είχε καταναλώσει αλκοόλ, αν είχε καταναλώσει ναρκωτικέ ουσίε, ποια ήταν η συμπεριφορά του, ποια ήταν η συμπεριφορά των άλλων. Έτσι λοιπόν μπορούμε να φτάσουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Οι ειδικοί οδική ασφάλεια θα σα έλεγαν, αν του ρωτούσατε, ότι χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία. Βρισκόμαστε στη συζήτηση με τον κλάδο, με διάφορα εμπλεκόμενα μέρη. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το κόστο πρώτον και το δεύτερο, πώ μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτά τα terabyte δεδομένων και να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά. Η κυρία Γκαρσία τώρα. Συμφωνώ με εσά. Το ιδανικό σενάριο θα ήταν το μηδενικό. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε και για το όραμα 0, το Vision Zero. Αν ρωτήσετε τους πολίτες ποιος είναι ο σωστός αριθμός θανάτων στο δρόμο, η απάντηση θα είναι φυσικά ένας αριθμός χαμηλότερος από αυτόν που έχουμε. Αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής, εμείς θέλουμε να, υπάρχει, να υπάρχουν μηδενικοί θάνατοι. Κανείς δεν θα ήθελε κάποιο συγγενής του ή κάποιο κοντινό του άτομο να χάσει τη ζωή του στον δρόμο. Αναφέρατε καλές ιδέες για την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στο αυτοκίνητο. Νομίζω ότι σε όλα τα κράτη-μέλη δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγεί. σε κάποια κράτη-μέλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί το hands-free για τις κλήσεις, αλλά η ιδέα σας μου φάνηκε πολύ καλή. Τώρα, ο κύριος Ρικέ και άλλοι ανέφεραν ε, το ζήτημα των θανάτων ανά, ανά χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί. Πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε τα στοιχεία. Η Γαλλία έχει κάνει βήματα σε αυτό το τομέα και θα πρέπει επίσης να ε, μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον κατάλληλο δίκτυο ώστε να ξέρουμε πόσα χιλιόμετρα έχουν διανυθεί. Παρ' όλα αυτά, δεν θα πρέπει να λέμε ότι η θάνατη ανά χιλιόμετρα είναι το κατάλληλο μέτρο και ο κατάλληλος δείκτης. Αν διανύαμε 10% παραπάνω χιλιόμετρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θάνατοι μειώνονταν κατά 5% θα λέγαμε τα καταφέραμε. Αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό το 5% είναι κάτι το θετικό. Η μόνη σωστή μέτρηση είναι η θάνατη ένα εκατομμύρια του πληθυσμού. Οι Αμερικάνοι στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν, ε, ε, ε, χρησιμοποιούν το πώς είναι η θάνατοι ανά όχημα και ανά τα οχήματα που υπάρχουν. Ούτε αυτό το θεωρώ σωστό. Ο κύριος Ρικέ ανέφερε και άλλα σημαντικά ζητήματα όπου στην ουσία περιγράφεται το ασφαλές σύστημα. Ναι, η, η συμπεριφορά του, οδού είναι οδηγού συγγνώμη, είναι ιδιαίτερα σημαντική, αλλά και η κατάσταση του οδοστρώματος. Θέλουμε ένα σύστημα το οποίο μπορεί να προβλέπει και να μειώνει τα λάθη έτσι ώστε να μην χάνουν τη ζωή τους οι άνθρωποι. κυρία Ντεπαρνέ αναφέρθηκε στα όρια ταχύτητας και το ποια είναι η κατάσταση στην Ευρώπη που υπάρχει κατακαιρματισμός. Πρόκειται για αρμοδιότητα των κρατών μελών και φυσικά υπάρχουν ε, όρια 130 στη Γερμανία, 140 στη Βουλγαρία, 140 στην ε, Πολωνία, στο Βέλγιο, επίσης 140 στην Εστονία το ανώτερο όριο είναι 100 και η Ολλανδία έχει μειώσει το όριο στα 100 κατά τη διάρκεια Δεν είστε οι πρώτοι που μου αναφέρετε ότι θα πρέπει να κάνουμε μια τέτοια σύσταση. Στόχος είναι βέβαια να δημιουργήσουμε μια προστιθέμενη αξία. Χρειαζόμαστε γνώμες ε, ειδικών εμπειρογνωμόνων στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Και πολύ σωστά αναφερθήκατε στη σύνδεση με την Πράσινη Συμφωνία. Δηλαδή ότι θα πρέπει παράλληλα να φροντίσουμε και για τη μείωση των εκπομπών και για τη βελτίωση του ε, αέρα. Μπορώ να συνεχίσω λίγο ακόμα. Έχετε ένα λεπτό. Θα ερευνήσουμε τις ε, προεκτάσεις που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των αυτόματων οχημάτων επίσης. Το ζήτημα των μοτοσυκλετιστών και η ασφάλεια των μοτοσυκλετιστών. Ο κύριος Βαντεκάμπ είναι εκεί πίσω και παρακολουθεί αυτή την απάντηση. οι ευάλωτοι χρήστε ε, τη οδού συμπεριλαμβάνουν και τους μοτοσυκλετιστέ. Αναφέρατε πάρα πολύ σωστά τα προβλήματα. Ότι υπάρχουν δηλαδή προβλήματα υποδομών. Ο ατομικός εξοπλισμό ασφαλεία είναι υποχρεωτικός και υπάρχουν πολύ αυστηρά μέτρα σε κάποιες χώρες όπως η Γαλλία. Σε κάποιες περιπτώσει υπάρχουν και απαλλαγέ και βοηθήματα για την αγορά αυτού του εξοπλισμού από τους οδηγούς. Αναφέρατε επίσης την εκπαίδευση και το πόσο, το σημαντικό είναι οι χρήστες να χρησιμοποιούν σωστά το οδικό δίκτυο. Η κυρία Γκραπίνη είπε κάτι με το οποίο συμφωνώ. Μιλήσαμε για τη μικροκινητικότητα, για τα πατίνια. Δεν έχουμε ακόμα αρκετά στοιχεία για αυτά τα οχήματα. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Φυσικά έχουν αναφερθεί αρκετά μεμονωμένα προβλήματα. Η κυρία ε, Τάξ αναφέρθηκε στο το κατά πόσον θα μπορέσει να υπάρξει ένας οργανισμός για την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη. Υπάρχουν κάποια ζητήματα προϋπολογισμού που προκύπτουν για τη δημιουργία νέων οργάνων και υπηρεσιών. Όμως θα πρέπει να δούμε και κάτι άλλο σε σχέση με την συλλογή δεδομένων. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε ε, και είναι μια καλή ιδέα και θα βοηθήσει τη συλλογή δεδομένων. Προς τον κύριο Λούκεν. Έχω απαντήσει ήδη στην ερώτησή σας. Γίνονται διάφορες συστάσεις στα κράτη-μέλη και αυτό είναι μέρος της δουλειάς μας. Δίνουμε συστάσεις. Εγώ ωστόσο δεν θέλω να θεωρηθώ ένας ειδήμονας που γνωρίζω τα πάντα για την οδική ασφάλεια και επιβάλλω συστάσεις στα κράτη-μέλη. Στόχος είναι να ανταλλάξουμε απόψεις, να κάνουμε προτάσεις και με βάση αυτούς τους νέους δείκτες επίδοσης, τους KPI, θα έχουμε μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων. Τώρα για τα Segway και τα πατίνια. Θα πρέπει να δούμε ποιες μετακινήσεις αντικαθιστούν. Αν δηλαδή κάποιος δεν χρησιμοποιεί πια το αυτοκίνητο και χρησιμοποιεί ένα πατίνι, τότε ίσως υπάρχει κάποια βελτίωση. Αν όμως σταματάει να χρησιμοποιεί το λεωφορείο ή το ποδήλατο και παίρνει το πατίνι, τότε δεν κερδίζουμε κάτι. Δημιουργείται μια νέα κατηγορία οχήματος με πολύ μικρές ρόδες, με προβλήματα ισορροπίας και αυτό δημιουργεί και ζητήματα ασφάλειας. Υπάρχει μία έρευνα ε, η οποία αυτή τη στιγμή διεξάγεται σε αυτό το τομέα. Αξίζει λοιπόν να σκεφτούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, ε, κοινέ κατευθυντήριες γραμμές για την χρήση αυτών των μεθόδων μικροκινητικότητας. Κυρία Ντέλη, μιλήσατε τελευταία και δεν έχω πολύ χρόνο να σας απαντήσω. Αναφερθήκατε στην ταχύτητα και για τα οχήματα SUV. Πρόσφατα αξιολογήσαμε αυτό το ζήτημα. Οι θάνατοι μεταξύ ποδηλατών και πεζών μειώνονται πολύ, με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα σε σχέση με θανάτους ατόμων που βρίσκονται μέσα σε αυτοκίνητα. Ε, τα στοιχεία είναι τραγικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάποιοι αναφέρουν ότι αυτό οφείλεται στην αυξημένη αγορά SUV. Μία μελέτη που έγινε για το Κοινοβούλιο δεν κατέδειξε οριστικά στοιχεία, σε οριστικά στοιχεία σε σχέση με το κατά πόσον τα βαρέα, πιο βαρέα οχήματα οδηγούν σε περισσότερους θανάτους ευάλωτων χρηστών του δρόμου. Και επίσης έχουμε θέμα ορισμού. Τι είναι το SUV, Υπάρχουν μικρά οχήματα SUV και τεράστια οχήματα SUV. Θα πρέπει να το ορίσουμε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, όσο μεγαλύτερο και πιο βαρύ είναι το όχημα, τόσο περισσότερε είναι και οι εκπομπέ μέσα στι πόλει. Δεν λέμε βέβαια ότι θα επιβάλλουμε κάποια ρύθμιση σε σχέση με τα οχήματα SUV, αλλά ότι αυτό πρέπει να το μελετήσουμε περαιτέρω. Ζητώ συγγνώμη που ε, αν δεν έχω απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις ε, και χάρηκα πολύ που συζήτησα μαζί σας. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Baldwin για το σύνολο των απαντήσεών σας. Μιλήσατε αρκετά το χρόνο το θέμα της οδικής ασφάλειας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και νομοθέτες και τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί δεν αρκεί να κάνουμε μεγάλες συνόδους κορυφής στο και ούτω καθεξής για να προωθήσουμε την προτεραιότητα αυτή, γιατί το είπατε, Μία ζωή που σώζεται είναι μια ζωή που σώζεται και οποιοδήποτε στιγμή μπορεί να συμβεί ένα δράμα, μπορεί να λέμε ε, ναι η ταχύτητα ή το άλλο, το ένα ή το άλλο θα πρέπει να ενισχύσουμε ωστόσο την ασφάλεια στους δρόμους μας. Μπορούμε να ευχαριστήσουμε, να χειροκροτήσουμε νομίζω τον κύριο Μπόλτουιν, πάντοτε μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε κοντά μας και πολύ ε, θα παρακολουθήσουμε και θα σας τροφοδοτήσουμε γιατί θα πρέπει πραγματικά να ασχοληθούμε πολύ σοβαρά με αυτό το θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνει η συνεδρίασή μας. Ε, ναι, όλα τελειώνουν. Δεν θα είμαι αύριο το πρωί εδώ. Θα έχω τη χαρά και την τιμή να αντικατασταθώ από τον συνάδελφο Έτχεν, που τον ευχαριστώ και τον προτέλω. Να μην ανησυχείτε. Αύριο το απόγευμα επανέρχομαι δρυμύτερη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα στη συνεδρίαση.